Monsieur le candidat Κύριε ψήφο επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, καταρχήν ζητώ από τον τύπο να αποχωρήσει. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας θυμίζω ότι ο υποψήφιος επίτροπος θα είναι στη διάθεση του τύπου μετά την ακρόαση. Ας αρχίσουμε. βρισκόμαστε υπό, υπό αυστηρή χρονική πίεση. Ο υποψήφιος κύριος Λεβαντόφσκι δικαιούται τρεις ώρες χρόνο. Ούτε ένα λεπτό λιγότερο, αλλά ούτε και ένα λεπτό περισσότερο. Διότι μετά πρέπει να εκενώσουμε την αίθουσα για να την αφήσουμε ελεύθερη για μια επόμενη ακρόαση. Αυτή εδώ η ακρόση μεταδίδεται άμεσα μέσω του ίντερνετ διαδικτύου. Είναι δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και οι δημοσιογράφοι και τα μέλη των άλλων θεσμικών οργάνων, οι διπλωμάτες είναι παρόντες, τους χαιρετίζω. Η συνεδρίασή μας αυτή γίνεται υπό την Προεδρία της Επιτροπής Προπολογισμών με τη βοήθεια της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προπολογισμού. Χαιρετίζω τον Πρόεδρο Λεμαγκίστρης και τα μέλη της Επιτροπής αυτής θα έχουν το δικαίωμα 35 λεπτά σε ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων με τον υποψήφιο. Η Επιτροπή Γεωργίας και η Περιφερειακή Επιτροπή επίσης εκλήθησαν και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο ίδιος ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής θα θέσει ερωτήσεις στο όνομα της επιτροπής του. Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννους Λεβαντόφσκι, υποψήφιος επίτροπος για τον οικονομικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό. Τον κύριο Λεβαντόφσκι τον γνωρίζουμε. Αλλά τον επίτροπο Λεβαντόφσκι δεν τον γνωρίζουμε, τον υποψήφιο επίτροπο εννοώ. Σύμφωνα λοιπόν με τις κατευθυντήρες γραμμές για την έγκριση για τις Κομισιόν, παράρτημα 17 του κανονισμού, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει τον υποψήφιο επίτροπο με βάση τις γενικές του δεξιότητες την δέσμευσή του υπέρ του ευρωπαϊκού οράματος και την προσωπική του ανεξαρτησία. Επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί η θέση του όσον αφορά το ενδεχόμενο χαρτοφυλάκιο που θα πάρει και την ικανότητα επικοινωνίας του. Σας θυμίζω ότι πριν την ακρόαση ο υποψήφιος απάντησε γραπτά σε ένα ερωτηματολόγιο οι γραπτές ερωτήσεις, απαντήσεις, συγγνώμη, οι γραπτές απαντήσεις που έχουν μοιραστεί σε όλες τις γλώσσες και υπάρχουν και έγγραφα το βιογραφικό σημείο του κ. Βανός, φυσικά ημερήσια διάταξη. Το βιογραφικό είναι στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Η δήλωση συμφερόντων του κ. Λεβαντόφσκη στα αγγλικά. Το mission statement, δηλαδή η αποστολή που το ανέθεσε ο πρόεδρος Μπαρόσο, το ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις και η επιστολή του Πρόεδρου Μπαρόσο. Τέλος, ειδού οι όροι με βάση του οποίου θα διεξαχθεί αυτή η συνεδρία και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων από τον υποψήφιο και από τα, τους συναδέλφους ευρωβουλευτές για το ότι ο χρόνος ομιλίας θα είναι πολύ περιορισμένος. Και είμαι υποχρεωμένος να έχω τον αχάριστο ρόλο να διακόπτω αυτούς οι οποίοι θα υπερβούν αυτό το χρόνο ομιλίας. Δέκα λεπτά για την εισαγωγική έκθεση του υποψηφίου επιτρόπου και ένα λεπτό μόνο για τους ερωτώντες με δυνατότητα απάντησης ένα λεπτό εκ μέρους του υποψηφίου και ένα δεύτερο δικαίωμα ερώτησης εκ μέρους αυτού που έθεσε την ερώτηση ή από άλλο μέλος της ίδιας ομάδας αν ο ερωτών δέχεται να εκχωρήσει το δικαίωμα απάντησης σε άλλο μέλος της ομάδας του. Εμείς στη γραμματεία θα τα σημειώνουμε όλα αυτά. Χρόνο μιλίας κατά ομάδα, κατά πολιτική ομάδα, έτσι ώστε να τηρηθούν οι κανόνες που εμείς ήδη ορίσαμε στους συντονιστές. Για, τον, για την κατανομή του χρόνου μιλίας. Ο κύριος Επίτροπος μας κάνει μια προφορική εισαγωγή 10 λεπτών. Μετά θα έχουν περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά ερωτήσεις. Μετά, αν μας μείνει λίγος χρόνος, θα σας προτείνω, κύριε Λεβαντόφσκι, να δευτερολογήσετε προκειμένου να κλείσει η συνεδρίαση. Ας ακούσουμε την εισαγωγική έκθεση του υποψηφίου επιτρόπου κυρίου Λεβαντόφσκι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάθεστε πίσω μου, σας έχω στην πλάτη μου, αλλά δεν φταίω εγώ για την διαρρυθμίση αυτή. Θα ήθελα να πω λίγα μονολόγια στη μητρική μου γλώσσα, τα πολωνικά, λίγα όμως μόνο. Γιατί στις δύσκολους καιρούς ε, η γλώσσα ήταν ένα εργαλείο για τη διατήρηση της ε, εθνικής ταυτότητας ε, και του εθνικού πολιτισμού και ανήκω σε μια γενιά που θυμάται τους αντίξους αυτούς χρόνους, ε, θυμάται το τίμημα της ελευθερίας και ε, την αξία της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα εγώ είμαι και υπέρμαχος της πολυγνωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο Λάσλο Σούριαν που βρίσκεται στην Ομίγυρη. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και ρεαλιστής, είμαι και πραγματιστής. Και για να διευκολύνω το έργο και των διερμηνέων και για να επιταχύνω και την ε, μεταξύ μας επικοινωνία θα συνεχίσω, λέει ο μιλητής, στα αγγλικά. Special to be... Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι στο παλιό γνωστό μέρος, αλλά με ένα νέο ρόλο. Είμαι επίσημα ακόμη ευρωβουλευτής και αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου εδώ, με τα παλιά μέλη της οικογένειάς μου και τα πολύ οικία μέλη, αλλά έχω ένα νέο ρόλο. Μάλιστα, κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στην Ομίγυρη και η Ντανούτα Χίμπνερ. Τώρα έχουμε ανάποδα, ανάποδα στους ρόλους, γιατί είναι τώρα πρόεδρος της, Επιτροπής, της Περιφερειακής Επιτροπής και έτοιμη να κάψει το νέο επίτροπο για τα θέματα αυτά. Έτσι οι, οι Πολωνοί συμβάλλουν και δίνουν νέα χρώματα και καινοτομούν στην διαδικασία έγκρισης. Βέβαια, έτσι μπορώ να αξιοποιήσω την προηγούμενη εμπειρία μου και να την χρησιμοποιήσω στην ε, μελλοντική μου αποστολή. Θυμάμαι όμως κάποιες εμπειρίες από όταν ήμουν ε, νεοεκλεγής Ευρωβουλευτής. Καθόμουν στο Προεδρείο και πίσω μου ο Μπέγκε, Μίλλερ και Βάλτερ. Και οι τρεις ήταν πολύ πιο έμπειροι από μένα. Αλλά ήταν και πολύ ενεκτική απέναντί μου και πολύ εξυπηρετικοί και με βοήθησαν. Γιατί ήμουν άπειρος τότε. Το ίδιο έκανε και ο συνάδελφος Σαλβαντόρ Καρίγα, ο Αλέλα Μασούρη, η κυρία Γκρέσλε, ο Τζέιμς Έλλης που ήταν τότε στην ομάδα μας. Και έκανε και μια δεύτερη ανακάλυψη τότε. Διαπίστωσα πως και οι άλλες ομάδες, ακόμη και οι ομάδες της αντιπολίτευσης, η αξέχαστη Κατρίν Κικέντ, η Γιούτα Χάουκ, η Αν Γένσεν, που θα μπορούσε να είναι υπόδειγμα να τη θέσουμε ως υπόδειγμα υπεύθυνη ε, πολιτικής συμπεριφοράς η Χέλγα Τρούμπελ. Είχαμε πολλές πολιτικές διαφωνίες μεταξύ μας, ε, εκπροσωπούμε διαφορετικές αξίες, αλλά όταν χρειάστηκε ενωθήκαμε για να προσπίσουμε μια κοινή θέση. Και αυτή ήταν η δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν τη ενώση. Και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέκτηνε τις αρμοδιότητες του και τις εξουσίες του και περιλήφθηκε τώρα στο πρωτογενές δίκαιο. Αυτή είναι και η αξία της ενότητας, η αρετή της ενότητας όποτε είναι απαραίτητη. Φυσικά υπάρχει και ένα αντίστοιχο αντιστάθμισμα στην πλευρά της Επιτροπής ε, που είναι ο συλλογικό χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Σώματο των Επιτρόπων. Και εγώ ασθενίζομαι πλήρω αυτή την αρχή, ότι εμεί είμαστε ένα επιτελείο, μια ομάδα που θα εξασφαλίσει τη συνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών και τη συνοχή του. Ο καθένα συμβάλλει με το δικό του τρόπο, αλλά όλοι μοιραζόμαστε τις ευθύνες και τις επομιζόμαστε από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση. Μερικές φορές μπορεί να είναι άβολο, αλλά σήμερα ε, καλό θα ήταν να αποφύγω βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ε, οριστικοποιηθεί η σύνθεση της Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη, όπως τις απαριθμό και στις γραπτές μου απαντήσεις. Η Επίτροπη έχουν ε, να αναλάβουν μία πλήρη ε, ημερήσια διάταξη και με πολλά αφιλεγόμενα και δύσκολα επίμαχα πολιτικά ζητήματα και μάλιστα αναλαμβάνει κάπως αργά το έργο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε να προσαρμοστούμε και στη νέα συνθήκη της Λισαβόνας. Τα βασικά μου συμπεράσματα είναι τα εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μείζον ε, ρυθμιστή, πολύ φιλόδοξο και προσπαθεί να επιβάλλει του κανόνε τη παντού, αλλά δεν έχει πάντα μεγάλη επιτυχία όπως συνέβη και στην Κοπεχάγη. Βέβαια, είναι σημαντική ρυθμιστική αρχή, αλλά τα δημοσιονομικά της μέσα είναι σχετικά περινυχρά. Μόνο το 1% του ΑΕΠ και 2% των συνολικών δημοσίων δαπανών. Δηλαδή, έχει περίπου ο κοινοτικός προϋπολογισμός της διαστάσεις του προϋπολογισμού της Αυστρίας και είναι ο μισός από τον προϋπολογισμό της ε, ε, Γαλλίας, ενώ αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα μόνο του γερμανικού προϋπολογισμού. Έχουμε λοιπόν σχετικά με τριοπαθή δημοσιονομικά μέσα και μάλιστα σε ένα πολυτάραχο κλίμα. Και μάλιστα δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διώκωσης του προπολογισμού μεσούσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης και του άγχους των κρατών μελών για τον προπολογισμό τους και τα προβλήματά τους. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς και με πενιχρούς πόρους καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα γεγονότα, τις αυξανόμενες μας ανάγκες, την υλοποίηση των πολιτικών μας δεσμεύσεων, που μερικές φορές αγνοούν τους, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Γι' αυτό και θα πρέπει να αναζητήσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στις τρέχουσες δημοσιονομικές προπτικές και καλύτερη αξιοποίηση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό κλάδο της σύμπραξης, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με άλλους οργανισμούς μετά την προσαρμογή στη Λισαβόνα θα πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη ημερήσια διάταξη και να τροποποιήσουμε τον προπολογισμό μας. Αυτό σημαίνει εξέλιξη για μένα και όχι επανάσταση. Καινοτομία δεν σημαίνει ε, παγίδευση στο παρελθόν, ούτε αγκύλωση στο παρελθόν. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, προηγούμενες ρυθμίσεις που τις έχουμε συσσωρεύσει χρόνο με το χρόνο, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε την αξία μας και να μην περιοριστούμε μόνο στους ίδιους πόρους, αλλά σε μια πολυεπίπεδη συνοχή που θα πρέπει να εδραιώσουμε. Επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε κάποια μορφή αρρωγής προς την Ήπεθρο, γιατί και η ανάπτυξη Ήπεθρο αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού μοντέλου. Σίγουρα η παράδοση δεν σημαίνει ότι είναι και παροχημένη και αναχρονιστική. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία θα πρέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός να γίνει πιο φιλικός προς το χρήστη αφενός. Αφετέρου όμως προσπαθούμε ε, να έχουμε θετικές δηλώσεις αξιοπιστίας για πρώτη φορά. Για να είναι λοιπόν φιλικός το χρήστη ο προπολογισμό και να στρέφεται προς τους πολίτες, θα πρέπει ε, να αποτελέσει μέλημα του Επιτρόπου και ο Επίτροπος θα πρέπει να αναβαθμίσει τη σχέση του όχι μόνο με τον κόσμο αλλά και με τους εκπροσώπους του λαού. Και οι εκπρόσωποι του λαού είστε εσείς οι ευρωβουλευτές. Και ευελπιστώ στο μέλλον με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και αμεσότητα να έχουμε καλές και αγαστές σχέσεις με, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά γιατί έχουμε και το τρίωρο σχεδόν της ακρόασης είμαι έτοιμο και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε προτινόμενε επίτροπε. Σας, σας συγχαίρω γιατί δεν εξαντλήσατε καν το δεκάλεπτο, μιλήσατε 8 λεπτά μόνο και έτσι θα δικαιούστε μια πιο εκτεταμένη δευτερολογία προς το τέλος της συνεδρίασής μας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων στους συντονιστές αρχής γενομένης από τον συντονιστή του ΕΛΚ, τον κύριο Σαλβαντόρ Γκαρίγκα. Έχετε το λόγο κύριε Γκαρίγκα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λεβαντόφσκι, αν υπάρχει ένα ιδεώδες προφίλ για τον υποψήφιο επίτροπο για τον προπολογισμό, σίγουρα είναι το δικό σα προφίλ, τα δικά σα χαρακτηριστικά. Γιατί έχετε πλούσια οικονομική και πολιτική πείρα, φτάσετε στι Βρυξέλλε ω παρατηρητή και μετά πλήρε μέλο αναλάβατε την Προεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμών κατά την ε, διαπραγμάτευση του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Έχετε άριστη γνώση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των περίπλοκων σχέσεών του με το Συμβούλιο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σας καθιστούν ιδεώδη υποψήφιο και είμαι βέβαιος ότι θα είστε σχεδόν ένας τέλειος επίτροπος. Έχω μια απλούστατη ερώτηση. Θα είστε ο πρώτο επίτροπος που θα εφαρμόσετε τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεράστια πρωτοβουλία σε δημοσιονομικά ζητήματα. Θα αξιοποιήσετε αυτή την πρωτοβουλία, ώστε να φέρετε τα δημοσιονομικά και θέματα προπολογισμού και τα χρηματοπιστωτικά στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων τη εκτελεστική επιτροπή. Απαντήσατε ότι θα, είστε ένα honest, honest broker στη σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία θα προωθήσετε κάποιον μηχανισμό μόνιμης διαβούλευσης και συνεννόησης με τους ε, συντάκτες των γνωμοδοτήσεων όπως είναι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, ο χρηματοπιστωτικός κανονισμός, ο δημοσιονομικός κανονισμός. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριος και απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σα. Φυσικά κανεί δεν είναι τέλειος. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη Λισαβόνα. Αυτό σημαίνει μεταβατικέ ρυθμίσει, που σε έναν βαθμό ήδη έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο συνδιαλλαγή το Νοέμβριο. Για τη συνεργασία τώρα με το Κοινοβούλιο υπάρχει η τυπική και η ουσιαστική πλευρά. Όσον αφορά την... το πνεύμα της συνεργασίας υπόσχεται πολλά. Όσον αφορά το τυπικό θα πρέπει να παραδιαπραγθούμε τη συμφωνία πλαίσιο, να την επικαιροποιήσουμε στο επίπεδο των νέων αυξημένων αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου και θα είμαι παρόν όποτε χρειάζεται και εδώ και σε άλλες αίθουσες του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό είναι στις κατευθυντήρες γραμμές του Πρόεδρου Μπαρόσο. Αναβάθμιση των σχέσεων με το Ευρωκοινοβούλιο. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις, μια από τις οποίες έχει ήδη γίνει από τον Οκτώβριο σε μια κρόση στο Κοινοβούλιο και θα απαντήσω φυσικά και στο αίτημά σας για πιο ουσιαστικέ και τυπικές ε, συναντήσεις μεταξύ μας. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπαγκαρίγκα δεν θα δευτερολογήσει. Ο κύριος Γκέραν Φέρμα. Ένα λεπτό. Κύριε Λεβαντόφσκι. Ο προπολογισμό δεν έχει μόνο νούμερα, έχει και πολιτικέ αξίε. Και πολλέ φορέ αμφιλέγεται αυτό όσον αφορά τι πολιτικέ κοινωνική συμπερίληψη, άνηση μεταχείριση, ισότητα των φύλων, οικογενειακό σχεδιασμό κλπ. Στον προπολογισμό του 2010, όπου θα έχουμε σύγκρουση αυτή τη κοινωνική συμπερίληψη και η μικροδιαχείριση δεν έχουν λυθεί μερικά θέματα. Το Συμβούλιο θέλει να το χρηματοδοτήσει περικόπτοντα το κύριο πρόγραμμα κοινωνική συμπεριληψη πρόγκρε. Ποια είναι η θέση σας κύριε Λεβαντόφσκι. Δεν θα πρέπει να έχουμε περισσότερε φιλοδοξίε στο πεδίο τη κοινωνική συμπερίληψη Και δεύτερον, για τη στρατηγική τη Λισαβόνα, Μερικοί κεντροδεξοί πολιτικοί θέλουν να στενέψουν του στόχου μόνο οικονομική ανάπτυξη. Να μην ασχολούμαστε με κοινωνικά θέματα. Ποια είναι η θέση σα εσεί όσον αφορά το πρόγραμμα του 2020 Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, για τις πολιτικέ πολιτικές της Ένωσης, οικονομικός προγραμματισμός και η αναπαραγωγική, αναπαραγωγική βοήθεια για τις γυναίκες. Ποια είναι η θέση σε αυτού κύριε Λεβαντόφσκι. Ο κύριος Λεβαντόφσκι έχει δύο λεπτά να απαντήσει για την κοινωνική συμπερίληψη. Μία αποκλεισμό. Αναφερθήκατε στο progress, ε, στο μέσον μικροχρηματοδότησης. Αυτό το μέσο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Κανένας δεν το αμφισβητεί προκειμένου να προωθηθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και να βρεθεί δουλειά για τους νέους. Αυτό που είναι επίδικο είναι από πού θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρω τη θέση του Κοινοβουλίου, αν θα είναι από το αποθυματικό ή όχι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αυξήθηκε όμω στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Αυτό το πέτυχε το Κοινοβούλιο να αυξηθεί ο φάκελο. Ξέρω όμω ότι σήμερα, επειδή τα περιθώρια είναι πολύ στενά, η πρόθεση είναι το Progress να μετατοπιστεί όσον αφορά στην Κομισιόν. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, δεν μπορώ να το πω, είναι κάπως πρόωρο. Πάντως, ε, νομίζω ότι είναι καλό εργαλείο η, το μέσο αυτό μικροχρηματοδότησης. Και φυσικά δεν η Λισαβόνα δεν αναφέρεται μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, εξίσου σημαντικές. Για πρώτη φορά με τη Λισαβόνα έχουμε την έννοια της γεωγραφικής συνοχής, όχι μόνο την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Μια νέα έννοια αυτή. Και χρειάζονται λεφτά και για αυτή τη διάσταση. Για την τελευταία ερώτηση για την ανάπτυξη δεν την κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Φέρμ πανέρχεται δευτερολογία. Στην ψηφοφορία που έχουμε στο Κοινοβούλιο για τον οικονομικό σχεδιασμό και θέματα ε, γεννητικής αναπαραγωγής. Ο προπολογισμό του 2010 έχει τροπολογία σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια ακριβώς για το θέμα αυτό οι τροπολογίες θα εμποδίσουν την Ένωση να υποστηρίξει προγράμματα οικονομικού σχεδιασμού με πληροφορίες για εκτρώσεις και οικονομικά μέτρα για την αύξηση της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών και εσείς ψηφίσατε υπέρ των περιορισμών αυτών παρά το ότι η Ένωση έχει δηλώσει ότι η καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία είναι αναγκαία αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Έχουμε και μια έκθεση για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβή, ίσης αμοιβή ανδρών γυναικών 2008. Έχουμε την έκθεση Μπότιγκεμ. Καταψηφίσετε το να ληφθούν νομικά μέτρα σε θέματα άνηση μεταχείριση θέματα μισθών. Και στην Φόντ Μπογκότιμαν ψηφίστε να απορριφθεί η νομική πρόταση για ίση μεταχείριση άσχετα με θρήσκευμα ή φύλλο ή γενετήσιο προσανατολισμό. Και ρωτώ, σε σχέση με αυτά τα θέματα άγγιση μεταχείριση, τα δικαιώματα των γυναικών εκτρώσεις, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, ποια είναι η θέση σας. Ένα λεπτό κύριο Λεβαντόφσκι. Αναγνωρίζω πλήρω την ευαισθησία που έχει αυτό το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και ορθά υπενθυμίσατε τον τρόπο που ψήφισα. Γιατί ψήφισα ε, στα πλαίσια της δικής μου πολιτικής οικογένειας και έχουμε κάποια δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των αναγκών του αναπτυσσόμενου κόσμου και ΥΟΣ δίνουμε 10 δισεκατομμύρια ε, ευρώ για την αναπτυσσόμενο κόσμο. Είμαστε οι πιο φιλάνθρωποι κατά κάποιο τρόπο, ο πιο φιλάνθρωπος ε, οργανισμός. Τώρα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε την ισότητα με τα δημοσιονομικά μέσα. Δεν είμαι κάπως πιο σκεπτικιστής τα θέματα ισότητα, ισότητα των φίλων, ισότητα ευκαιριών και όλα άλλα, τα άλλα που αναφέρατε μπορούν να ε, διαθετηθούν και με δημοσιονομικά μέσα. Και έχετε δίκιο ότι είχα μια συγκεκριμένη ψήφο ε, παρόμοια αυτή τη πολιτική μου οικογένεια για όλα αυτά τα θέματα. Για τη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γένσεν. Σας ευχαριστώ. Έχω υψηλέ προσδοκίε ε, από τον προτινόμενο επίτροπο που θα έχει πολύ δύσκολο έργο γιατί τον περιμένει η διάμεση αναθεώρηση και η επεξεργασία των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Και ένα από τα θέματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαμηλή επιρροή είναι το θέμα των εισοδημάτων, των εσόδων που αναφέρατε και σα ακροθυγώ. Το θέμα αυτό είναι πολύ περίπλοκο και έχει διάφορα rebates και οι διάφοροι πρόεδροι των επιτροπών προσπάθησαν να υποβάλουν προτάσεις χρήσιμες για αυτές τις επιταγές προς τα κράτη-μέλη και δεν ξέρω, είστε έτοιμος εσείς για μια εμβριθή και διεξοδική συζήτηση για το θέμα αυτό και ποιες είναι οι απόψεις, το όραμά σας για το πώς θα διαθετηθεί η πρόταση αυτή από τους ίδιους πόρους. Σας ευχαριστώ κυρία Γένσεν για τον, υπενιγμό, τον ευγενικό σας υπενιγμό. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Λεβαντόφσκι. Από ό,τι θυμάμαι, ο πρόεδρος είχε πρόβλημα όταν αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή φορολογία και τότε ήταν ίσως ε, το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη για ένα τέτοιο είδος φορολογίας και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποβεί εις βάρος του δεσμού της Ευρώπης με τον πολίτη, σε αντίθεση με όσα πιστεύουν ορισμένοι. Πάντως, όλο αυτό το έργο που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλη αυτή η προεργασία που έγινε και το θέμα της αναθεώρησης, γιατί η αναθεώρηση θα αγγίξει όλες τις πτυχές, ακόμη και τους ίδιους πόρους. Είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε μια νέα πρόταση για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, προκειμένου να γίνει σωστά αυτό το έργο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις εκθέσεις του Αλέλα Μασούρ. Γιατί εκεί έγιναν ειλικρινείς προσπάθειες, ε, ε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, προκειμένου να διευρυνθεί η συζήτηση. Είναι εύκολο να βρεθούν αδυναμίες ε, στις υπάρχουσες συμφωνίες. Γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων, διάφορες αντιφατικές διατάξεις και ούτω καθεξής. Τα λέω αυτά όλα στα γαλλικά για να αποτύσω φόρο τιμή και στον πρόεδρό μα. Είναι εύκολο να γίνει μια διάγνωση, αλλά πολύ πιο δύσκολο είναι να βρεθεί μια λογική λύση. Και λέω λογική, ορθολογική λύση, γιατί απαιτείται ομοφωνία και υπάρχει και το θέμα τη εθνική κυριαρχία. Γι' αυτό και θα πρέπει η λύση που θα βρεθεί να είναι πολιτικώ εφικτή. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για ένα αμυγό φορολογικό σύστημα στου ιδίου πόρου γιατί κάτι τέτοιο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ε, της πολιτικής ε, σκοπιμότητας εφικτότητας. Ίσως θα μπορούσαμε, ε, όπως πρότειναν εκθέσει του Κοινοβουλίου, να προχωρήσουμε σε δύο φάσεις, σε δύο στάδια. Γιατί στα έγγραφα αυτά, στις εκθέσεις του Αλέλα Μασούρ, βρίσκουμε τι είναι εφικτό προς το παρόν. Και για την αναθεώρηση και για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Η κυρία Γιάννησεν για ένα λεπτό. γνωρίζουμε ότι η συζήτηση αυτή θα συνδυαστεί με την ε, συζήτηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και γίνεται λόγος για αλλαγή της ε, ε κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, που θα λαμβάνει περισσότερη υπόψη το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την ευημερία των ζώων. Πρόκειται να εκπονηθούν κάποιες μελέτες για το θέμα αυτό, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαμε να έχουμε, είχαμε δει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στο προπολογισμό του 2009 προκειμένου να γίνουν έρευνες και προς του αυτούς. Τίποτα όμω δεν έγινε τελικά. Εσείς ως Επίτροπος θα μεριμνήσετε για να εισακουστούν οι επιθυμίες της Δημοσιονομικής Αρχής και να εφαρμοστεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Για ένα λεπτό, κύριε Λεβαντόφσκι. Φυσικά τρέφω τόσο σεβασμό προς το πρόσωπό σας που λέω ανεπιφύλακτα ναι, θα προωθήσω αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Και μάλιστα η κατάσταση αλλάζει. Δεν είναι το ίδιο τμήμα του προπολογισμού που είχαμε ε, προηγουμένως. Ήταν 70 με 80%, τώρα θα είναι 30-33%. Πάντως αυτός είναι ο τομέας που επικρίνεται περισσότερο από την κοινή πολιτική. Αυτό που θέλουμε τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και η προσωπική μου γνώση, είναι ότι δεν θέλουμε επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Γιατί κάτι τέτοιο θα θέσει τέρμα στην ε, κοινή γεωργική πολιτική. Εγώ έλεγα να ε, εφαρμόσουμε προαιρετική βάση, προαιρετική διαφοροποίηση, το modulation και να μπορούν προαιρετικά τα κράτη-μέλη να διοχετεύσουν τις γεωργικές ε, δαπάνες, τις γεωργικές ενισχύσεις προς τους διάφορους τομείς, προκειμένου να διαφυλάξουμε και την υπεθρό και την αγροτική οικονομία. Πάντως η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του προβλήματος και των επικρίσεων που συγκεντρώνει αυτό το τμήμα της κοινή ζωρικής πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Από τους πράσινους τώρα η κυρία Ντουιρόν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Λεβαντόφσκι. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την έκβαση των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Τότε οι κλιματικές αλλαγές θεωρούνταν από τους περισσότερους ως ύψιστη προτεραιότητα. Δεύτερη ήταν ανταγωνιστικότητα και ενέργεια. Σας ερωτώ, εστερνίζεσαι αυτές τις προτεραιότητες? Γιατί σε μερικές δηλώσεις που είχατε κάνει πριν σας προτείνουν για επίτροπο, δημιούργησα την εντύπωση ότι για εσά η ανταγωνιστικότητα είναι πιο σημαντική από τις κλιματικές αλλαγές. Μιλήσατε και για τη γεωργική πολιτική. Σας ερωτώ, γιατί απαντήσατε εν μέρη πριν στην ερώτηση. Πώς θα προσανατολίσετε τις ε, άμεσες ενισχύσεις, γιατί αναφερθήκατε στην προαιρετική βάση. Εγώ προτιμώ κάτι πιο δεσμευτικό και κυρίως ένα προσανατολισμό της γεωργίας προς την αηφόρο ανάπτυξη και μια πραγματική γεωργία με υποχρεωτική βάση. Για το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιταχύνει την ε, στρατηγική του 2020. Ποια η σχέση της στρατηγικής αυτής με το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Ο κ. Λεβαντόφσκι, δύο λεπτά απάντηση. Φυσικά συζητούμε το, το θέμα των κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη με πολύ διαφορετικό τοπίο που βλέπουμε στα παράθυρά μας σήμερα. Πάντως, ε, οι νέες δεσμεύσει θα οριστικοποιηθούν μετά την έκβαση της συνδιαλέγης. Πάντως, δεν μιλούμε μόνο για τα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το αίτημα των κρατών μελών. Μιλούμε για 150 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να βρεθούν από τον κοινό προπολογισμό. Και χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αύξησε τα οριζόντια προγράμματα κατά 50 εκατομμύρια για το 2010, έχουμε το 2010 υποέλεγχο πια. Το έχουμε θέσει υποέλεγχο. Τώρα αυτό που έπεται είναι να βρούμε ε, συμπληρωματικά κονδύλια για το 2011 και 2012. Και ο άγνωστος χ είναι πώς θα χρηματοδοτήσουμε την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών για το 2013 και μετά δεν ξέρω αν θα χρηματοδοτηθούν από τον κοινό προπολογισμό ή θα πρέπει να ιδρυθεί ένα αυτόνομο ταμείο κλίματος. Αυτή είναι όμως μια ερώτηση που θα απαντήσουμε στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, εγώ είμαι υπέρμαχος μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, και φυσικά θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ε, λαϊκή σοφία, στην τοπική σοφία. Και ο επαναπροσανατολισμός της γεωργικής πολιτικής περιλαμβάνει την ε, πολλαπλή διασταύρωση, την πολλαπλή συμμόρφωση, αλλά θέλουμε ένα καλύτερο προσανατολισμό, γιατί θα πρέπει να γίνει κάποια προσαρμογή και για τα νέα κράτη-μέλη και νομίζω ότι αυτή η λύση της προαιρετικής βάσης είναι καλύτερη. γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις νέες τεχνολογίες ε, και στις νέες χώρες για να έχουμε πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και γεωργία. Το 2020, πριν τη στρατηγική του 2020 θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση. Αυτή είναι η διασύνδεση μεταξύ τους. Οι προτεραιότητες ε, θα καθοριστούν όχι στο Ερεινό Συμβούλιο, αλλά στο Θερινό. Και θα δούμε ποια θα είναι η συμφωνία για τις πολιτικές προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντουρό, θέλετε να αναφερθώ, όχι κύριε Τρούπελ. Ναι, στη δεύτερη ερώτηση θα αναφερθώ, θα σας μιλήσω στα γερμανικά. Έχοντας ακούσει λιγάκι αυτά που είχατε να μας πει κύριε Λεβαντόσκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κατανοείτε κατ' ουσίαν το πολιτικό σας ηγετικό ρόλο ως Επιτρόπου σε όλα τα δημοσιονομικά αυτά θέματα. Είδαμε την αποτυχία της διάστησης Κοπενχάγης και ξέρουμε ότι και πολιτικά αλλά και ε, μέσα στα πλαίσια του προπολισμού πολλά πρέπει να τροποποιηθούν εάν θέλουμε καλύτερα και οικολογικά αποτελέσματα επόμενα χρόνια αλλά και οικονομικά μεγαλύτερη επιτυχία. Για να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε μια καλύτερη ουσιαστική κατανόηση των θεμάτων και τι θα γίνει μέσα στα πλαίσια της μεσόπροθεσμης δημοσιονομικής ε, πρόβλεψης ε, αυτή η κριτική στάση που εκπροσωπείται εδώ αυτή τη στιγμή είναι αυτό που χρειάζεται η Κομισιόν ή θα πρέπει να έχουμε μια ε, πιο ηγετική στάση, πιο ισχυρό ρόλο της Κομισιόν τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Λεβαντός και ένα λεπτό. Αυτό που μου αρέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι πολιτικές δεσμεύσει δεν χρηματοδοτούν επαρκώς. Αυτό έγινε όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τις κλιματολογικές αλλαγές και για τη διάσκεψη Κοπενχάγης. Γιατί τελικά οι πολιτικές ε, αποφάσεις δεν έφτασαν στις προσδοκίες ουδενός. Αυτή η πολιτική του 2020 προβλέπει περιβαλλοντικά προγράμματα στην Ευρώπη, αλλά σαν κύρια προτεραιότητα. Και αυτό όσον αφορά τη χρηματοδοτική διάσκεση, σημαίνει ότι θα πρέπει η προτεραιότητα αυτή να αντικατοπτρίσει στον προπολογισμό. Το πρόβλημα είναι ότι ε, δεν έχουμε πάρα πολύ αρκετό χρόνο μεταξύ της αναθεώρησης και το θα πρέπει να γίνει μετά τον Ιούνιο για τη στρατηγική αυτή του 2020. Γιατί αυτά τα θέματα, τα περιβαλλοντικά, τα κλιματολογικά, είναι η κύρια προτεραιότητα για το 2020. Και αυτό θα πρέπει βέβαια να έχει επιπτώσεις. Στην δημοσιονομική διάσκεψη, διάσταση, συγγνώμη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Για την ομάδα η σειρά, ο κύριος Μπόκος αποσιάζει. Ο κύριος Έπινγκ, θέλετε να πάρετε το λόγο, ένα λεπτό. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα υποβάλω την ερώτησή μου στα Ολλανδικά. Μα... Αναφέρομαι στο θέμα των δύο πόρων. Είπατε εσείς ότι καταρχήν είσαστε κάπως επιφυλακτικός. Δεν ε, παραμένετε υπερβολικά προσκολλημένος σε αυτό. Αλλά πώς σας φαίνεται η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Φόρου, ο κ. Δεχάν, ο κ. Φορσέντατ είναι υπέρμαχοι αυτών. Και λένε ότι θα είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, αν έχουμε ένα πράσινο, αν θέλετε, κάλυμα για αυτά. Αλλά πάντως πρόκειται για φορολογικό φόρο ευρωπαϊκό. Ο κ. Λεβαντός για δύο λεπτά. Έχουμε μόλις ολοκληρώσει μια μεγάλη αναθεώρηση χάρη στον μας και ξέρετε ότι μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ολλανδία και η Αυστρία είναι εκείνες που ασχολούνται με το θέμα του Ευρωπαϊκού φόρου κυρίως. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το θέμα της ομοφωνίας των αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα ιδιών πόρων. Θα πρέπει να υπάρξουν πολιτικά ε, λύσει υπάρχουν υποψήφοι για φορολογία και στις προτάσεις κ. Σάιερ του 2004 και έχουμε και άλλες προτάσεις επιτάπητος. Έχουμε μία ομάδα υποψηφίων για την φορολογία με αυτή την καινοτόμα πλευρά των εκπομπών οξυδίου του άνθρακα. Όλα αυτά θα πρέπει να εξαστούν κάτω από το πρίσμα της ε, απλής εφαρμοσιμότητας της ε, δυνατότητας της φορολογικής εφαρμογής. Εγώ δεν αποκλείω λοιπόν τις δύο ε, πόρους, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα προς την αρχική ιδέα και το πνεύμα της εθήκης της Ρώμης. Τώρα είμαστε αντίθετοι με την ιδέα του και το πνεύμα της συνθήκης Ρώμης στον αφορά του δύο πόρους. Σας ευχαριστώ κύριε Έπινγκ. Δεν θέλετε να θετρολογήσετε. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας είχε πει ότι τα χρήματα δεν έχουν οσμή. Non-OLED. Τώρα εμείς θα δούμε αν έχουν χρώμα τα χρήματα. Ο κύριος Μίγκελ Πόρτες για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επιτροπέ, η ερώτησή μου είναι η εξή. Σας άκουσα να μιλάτε για τους ιδίους πόρους ε, με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ε, την πρώτη φορά μας, είπε, μας είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ομοφωνία. Τη δεύτερη φορά είπατε ότι δεν αποκλείεται καμία λύση για την αύξηση των ιδίων πόρων. Και την τρίτη φορά ιδιαίτερα για τη δυνατότητα της φορολογίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είπατε ότι ίσως κάτι τέτοιο βλάψει την οικονομία. Για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ξέρω ότι και από τη δική σας πολιτική οικογένεια πολλοί πρωθυπουργοί και μάλιστα ιδιαίτερα ο κύριος Σαρκοζή και ο Γκόρντον Μπράουν από άλλη πολιτική οικογένεια έκαναν δηλώσεις υπέρ της φορολογίας αυτής των οικονομικών συναλλαγών. Ερωτώ λοιπόν, γιατί μια και άλλαξε η θέση πολλών πρωθυπουργών και μάλιστα σημαντικών, γιατί εσείς εμένετε σε μια θέση αντίθετη με τη φορολόγηση αυτή. Γιατί δεν νομίζω να οφείλεται αυτό στην ομοφωνία, μάλλον στη δική σας προσωπική γνώμη θα οφείλεται αυτή η στάση σας και η αιμονή σας. Ευχαριστώ, δύο λεπτά Λεβαντόφσκι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτός και ελπίζω να παραμείνω ανοιχτός όσον αφορά τα θέματα και της Επιτροπής παραπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά η ιδέα θα πρέπει να περί κάποια κριτήρια. Ξέρω ότι εκτός από τους υποψήφους αυτούς για τους φόρους, οι δυναμοσυνομικές, οι χρηματοπιστικές συναλλαγές είναι και μια επιλογή που υπάρχει επιτάπτως. Από όσο ξέρω και στο ε, πρόσφατα απέφυγε να υποστηρίξει. Αλλά είναι και αυτό ένα από τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχει επιτάπητος. Σαν παραδείγματος χάρη μια από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εγώ είμαι ανοιχτό στην ε, εξέταση για να καταλήξουμε σε κάποιο τολικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις προτεραιότητες που αναφέρονται στη στρατηγική του 2020 και κατόπιν είμαστε υποχρεωμένοι να προτείνουμε διαφορετικές μεθόδους, όχι συνοχή του συστήματος ιδιών πόρων. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005. Τα κριτήρια όμως είναι πολύ απλά. Απλότητα, ουδετερότητα φορολογική, διαφάνεια και χαμηλό κόστος συλλογής του φόρου αυτού. Και εγώ παραμένω προς κολλημένο σε αυτή την στάση. Είμαι ανοιχτό σε την πρόταση υποψηφίων για νέους σπόρους, για νέους ιδίους σπόρους που έχουν ήδη υποβληθεί. Υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα think tank γύρω από τα ευρωπαϊκά σώματα που δεν είναι απόλυτα για ποια κριτήρια θα ε, υιοθετούν. Ευχαριστώ κύριε Σπόρτας. Ένα λεπτό. Δεύτερη ερώτηση για το θέμα της συνοχής. Όχι μόνο της εδαφικής, αλλά και της κοινωνικής. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η εδαφική συνοχή είναι σημαντική και για την κοινωνική συνοχή. Αλλά δεν αρκεί. Δεν έχουμε σημαντικές πολιτικές για την κοινωνική συνοχή. Σας ερωτώ λοιπόν. Θα ήσταν έτοιμος να εξετάσετε στα πλαίσια της αναθεώρησης των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών και να εξετάσετε τη δυνατότητα σύσταση ενό συμπληρωματικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για να συμπληρώνουν τα συστήματα κοινωνική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και τα πιο αδύναμα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριε Λεβαντόφσκι. Κοιτάξτε, η θέση μου μέχρι τώρα είναι να σέβομαι τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποια προβλήματα και με διάφορες εξωτερικές υπηρεσίες και διάφορα εξωτερικά και α, ανεξάρτητα ταμεία που υπάρχουν, ε, παραδείγματος χαρακτηριστικό ταμείο ανάπτυξη. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Πώ θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τι κρεματολογικέ αλληλεγγύε με ένα ειδικό ταμείο ή σαν να είναι μέσα στα πλαίσια του κανονικού κοινοτικού προπολισμού. Η στάση μου είναι να σέβομαι τις μέχρι τούδε συμφωνίες. και να μην ε, ξεχνάμε αυτά τα εξωτερικά μέσα που υπάρχουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυξάνονται και πληθύνονται πάρα πολλά μέσα εκτός του προπολογισμού και αυτόν τον τρόπο χάνουμε τη δυνατότητα ελέγχου και αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού τη δυνατότητα για τις δαπάνες αυτές. Αυτή είναι η σημερινή μου θέση. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ. Κανονικά θα έπρεπε να μιλήσει εκπρόσωπος του ΕΦΤ, αλλά η κυρία Μάρα Αντρέασεν δεν είναι εδώ, ο κύριος Μουργαντή, ούτε και εκείνος. Μία γραμμένη. κυρία Βέρτμαν, μου είπε ότι δεν θα μπορούσε να είναι παρούσα. Ζήτησε γνώμη για την αποσίαση, γιατί είχε δυσκολίε μετάβαση. Ο κύριο Φαντερ Στόμπ αποσιάζει επίση. Λοιπόν, προτείνω να δώσουμε το λόγο στην κυρία Χολμάιερ για να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα απάντηση του κυρίου Καρίκα που δεν χρησιμοποιήσει. Δύο λεπτά κυρία Χολμάιερ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θα σας την εξή ερώτηση όσον αφορά την πολιτική των κτηρίων. Κατά πόσο ο νέος Επίτροπος προτίθεται να ενημερώνετε έγκαιρα την ε, Επιτροπή Προεπισμών για νέα σχέδια και να μας εμπλέξετε στην ε, φάση της προετοιμασίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ε, καθυστερήσεις. Και επίσης θα δώσετε στην Επιτροπή Προεπισμών μια γενική εικόνα των υπαρχών οκτηρίων και των αναγκών για το μέλλον και μια κλίδα της πολιτικής για το κτηρίων για το μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική αυτή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Λεβαντόφης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτό είναι μια δήλωση μέσα στα πλαίσια της ε, διαβούλευσης του Νοεμβρίου. Η συμφωνία πάνω σε ένα μακρόχρονο όραμα της πολιτικής κτηρίων με ένα όραμα που ε, καταστρέφει το λόγο του ότι υπήρχαν αγορές από εδώ και από εκεί και μέσα στα πλαίσια μιας αίτησης μεταφοράς ε, κονδυλίων που έφτανε τελευταία στιγμή στα χέρια του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο την συνέργεια μεταξύ της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων όταν αγοράζουμε κάτι στο εξωτερικό σε χώρες εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα παλαιό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί προτιμούμε να αγοράσουμε παρά να νοικιάσουμε. Και τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να εντεχθούν μέσα στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής. Και εγώ θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το, στη συνολική εικόνα των κτηρίων που έχουν ε, αγοριστεί από τα άλλα θεσμικά όργανα. Euh, Τώρα θα περάσουμε στι ερωτήσει Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. 35 λεπτά. Θα παραχωρήσω την Προεδρία και το Σφυράκι στον κύριο Ντεμάγκιστρη, Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, χαιρετίζω και χαιρετίζω και τον υποψήφιο επίτροπο κ. Λεβαντόφσκι. Πριν όμως δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες ελέγχου του προπολογισμού για το χρόνο που έχουμε, θα ήθελα να παρουσιάσω ορισμένα θέματα ως πρόεδρος. Διάβασα με πολύ προσοχή αυτό που γράψατε και θα ήθελα με διευκρινήσει προ το πώ σκοπεύετε, κύριε Επίτροπε, να πετύχετε ισορροπία ανάμεσα στην απλοποίηση από τη μία μεριά για να έχουμε πιο αποτελεσματικό ε, τρόπο χρήση των κονδυλίων και του κανόνε που χρειάζονται για να μην έχουμε ε, απάτε και μεγάλα λάθη. Δηλαδή, πώ θα απλοποιήσετε χωρί να καταργήσετε κανόνε οι οποίοι ε, εμποδίζουν τι απάτε και πώς σκοπεύετε να παρέμβετε στο λεγόμενο κίνδυνο του ανεκτού λάθος. Με ακρίβεια διάβασα ότι σκοπεύετε ότι θα συνεχίσετε τη γραμμή της δημοσιοποίησης των δικαιούχων των κοινωνικών κονδυνίων. Σκοπεύετε να αναφέρετε και αυτούς και τα κράτη που κάνουν παραβιάσεις και τι σκοπεύετε να κάνετε σε σχέση με τα κράτη που κατ' επανάληψη είναι υπεύθυνα για παραβίαση όσον αφορά τη χρήση κονδυλίων που δίδει η Ένωση. Εγώ, oh, Ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Η απλοποίηση δημοσιονομικών κανόνων είναι το πιο σύνθετο πράγμα. Από ό,τι ξέρετε, το ξέρουν τώρα οι συνάδελφοι Γκρέσλε και άλλοι, ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός 2002 ήταν υπεραντίδραση στην, κατα... στην κίνηση κατά της Επιτροπής Σαντέρ. Μετά είχαμε μια έκτακτη προσπάθεια απλοποίησης, να είναι πιο φιλική ως προς το χρήστη. Και το 2006 ε, ξεκίνησε και εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2007. Πρόκειται για τον τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και η Κομισιόν έχει φιλόδοξους στόχους. Θέλει να έχει μέσα και την έννοια του ανεκτού, του κινδύνου ανεκτού λάθους, αλλά και νέα εργαλεία μόχλευσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ιδιωτικέ και δημόσιε εταιρικέ σχέσει. Όσον αφορά το, τον ανεκτό κίνδυνο λάθους αυτή είναι μια έννοια που ξεκίνησε από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να την αναλύσουμε για να λαμβάνουμε υπόψη την σύνθετη φύση πολλών και διαφορετικών πολιτικών. Στην αρχή έχουμε την έρευνα. Οι πιο πολλές καταγγελίες προέρχονται από εκεί. Νομίζω η έρευνα και οι μεταφορές είναι οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι. Μετά θα έρθουν οι άλλοι τομεί. Μετά πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ της κόκκινης γραμμής 2% και τις διάφορες πολιτικές. Αυτό αναφέρεται στις παραγράφους και τα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού που έχουμε. Άλλο αυτό και άλλο η προσαρμογή στη Λισαβόνα. για να γίνει πιο φιλικό για το χρήστη ο δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά επαναλαμβάνω η Κομισιόν έχει φιλόδοξου στόχου ήδη από το 2005. Να έχουμε την θετικό DAS όσο πιο γρήγορα γίνεται. Declaration of Assurance όπως το λέμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και το λόγο στον κύριο Ήταλα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κύριε Λεβαντόφσκι, ήθελα να σας ρωτήσω για τα διορθωτικά ταμεία. Η χρηματοδότηση για τα διορθωτικά ταμεία, το 11% τουλάχιστον, είναι παράτυπη δαπάνη. Δηλαδή ο προπολογισμό στο σημείο αυτό δεν είναι αποδοτικός, δεν λειτουργεί σωστά. Έχουμε ένα σωρό παρατυπίε και αυτό αφορά περισσότερο από μία χώρε μέλη. Δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση του προγράμματο δράση για τα διευθυντικά ταμεία, ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα. Και μπορεί κανεί να αμφιβάλλει θεμετά. Είναι σωστό το action plan, λειτουργεί σωστά. Τι θα κάνετε έτσι ώστε όλε οι παρατυπίε αυτέ να ληφθούν πιο καλά υπόψη και τα λεφτά να χρησιμοποιούνται πιο σωστά και πιο αποδοτικά. Απάντηση. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Το 11% δεν είναι ανεκτό ποσοστό λάθος. Και αυτή είναι η αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής. Όμως, είχαμε και βελτιώσεις. Μεταξύ του 2004 και του 2008 και η διαδικασία απαλλαγής του 2008 το δείχνει αυτό. Αυτό το είπε και το ελεκτικό συνέδριο και είχαμε και μείωση του συνολικού όγκου λαθών στην εκτέλεση του προπολογισμού. Ξέρετε και όλοι ξέρουμε ότι το πρόβλημα με τη συνοχή είναι ότι το 80% το διαχειρίζεται τα κράτη-μέλη. σε πολλά επίπεδα. Ο φιλόδοξος στόχος να έχουμε την ε, βεβαίωση αυτή από τους ελεγκτές με πιστοποιητικό σε όλη την Ένωση, αυτό δεν το έχουμε πετύχει ακόμα και ότι και είναι ρεαλιστικό να ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε σχετικά σύντομα. Έχουμε διαφορετικές προδιαγραφές. Έχουμε πολλές χώρες μέλη. Δεν είναι εύκολο να πω ποια χώρα είναι να κατηγορηθούν. Θα μπορούμε βέβαια να αναφέρουμε τα ονόματα κρατών που καθυστερούν όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Αλλά δεν είναι καθόλου δημοφιλές αυτό στο Συμβούλιο ως μέθοδος. Οπότε δεν έχω πάρει ακόμη θέση. Γι' αυτό αναφέρθηκα στους δικαιούχους των κοινωτικών κονδυλίων. Γνωρίζω όμως το πρόβλημα των ομοσπονδιακών κρατών κυρίως. Σχετικά με το εθνικό DAS. Ο κύριος Ήταλα θα γίνει να δευτερολογήσει 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άλλο σημαντικό θέμα. Γεωργία. Στην έκθεση δραστηριότητα γενική Διεύθυνση Γεωργία είναι σαφέ ότι τα λάθη στην πολιτική για τη γεωργία του 2007 ήταν 1,58%. Στη Φιλανδία είναι 0,8%, στη Γερμανία 0,3%, στην Ισπανία 0,6% διαφορά. Σε άλλες χώρες το νούμερο είναι τελείως διαφορετικά. Βουλγαρία πάνω από 13%, Ρωμανία 12,5%, παρατυπίες εννοώ. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ελέγχων δεν λειτουργεί σωστά και οι κυρώσεις που επιβάλλει η Κομισιόν που θα μπορούσε να παγώσει κονδύλια ή να ανακτήσει κονδύλια, δεν φαίνεται ούτε αυτό να λειτουργεί. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ο κύριος Λιβαντόφσκι. Αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Στη μέθοδο αναφέρω ονομαστικά αυτούς που έχουν υποπέσει σε πτέσμα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι θέμα... Αναφέρεται χώρες όπου η παρατυπήση 0,3% η Γερμανία, Φερρυπίν. και άλλες που ξεπερνάνε το 10%. Η ερώτησή σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές αναχώρα. Αυτό ισχύει και για τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά για την ανάκτηση κονδυλιών, νομίζω έχουμε βελτίωση. Νομίζω ήταν 2,9 δις ευρώ πέρυσι. Καλό είναι το ποσό αυτό. Να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό που λέμε λάθος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι πάντα απάτη. Μπορεί να είναι ένα τυπικό λάθος και να μην είναι σπατάλι χρημάτων. Το λάθος δεν ισοδυναμεί με απάτη. Για μερικέ περιπτώσεις, στι οποίες ερεύνησε η Όλαφ, ισχύει αυτό, αλλά όχι σε όλες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σάφο Γκέιερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λεβαντόφσκι, κατά πόσο μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι η εξωτερική πολιτική της κοινότητας θα παραμείνει κοινοτική πολιτική και δεν θα είναι μια διακυβερνητική πολιτική στο μέλλον. Πώς προτείνετε να εξασφαλίσετε την δημοσιονομική διαφάνεια στον τομέα αυτό και να εμπλακεί πλήρω η νέα υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ζευμαντάφσκι έχει δύο λεπτά να απαντήσει. Η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Είναι το πιο εμφανές όργανο, θα έλεγα, μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης Λισαβόνα. Και είναι ένα όργανο sui generis, που διαχειρίζεται τους διοικητικούς τους πόρους και τις δικές της δαπάνες μόνη Το πραγματικό πρόβλημα τώρα για τον ελεγκτή είναι πώς, τι είδου ρύθμιση θα έχει για τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό για να δει τις λειτουργικές δαπάνες. Και το τμήμα προπολογισμό της Κομισιόν υπάρχει το διοικητικό σκέλος, όπως τα άλλα όργανα, αλλά να είναι υπόλογο, πλήρως υπόλογο έναντι του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Δηλαδή, όποια και να είναι η λύση, είτε αυστηρή διοικητική διαχείριση σου ή generis στην υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης, που θα πρέπει να συσταθεί μέχρι το τέλος Απριλίου, ή διοικητικές δαπάνες, όπως ορίζει η συνθήκη, ευθύνη της Κομισιόν. Και για τις δύο περιπτώσεις, την απαλλαγή τη δίνει το Κοινοβούλιο. Άρα είναι υπόλογοι πλήρως έναντι του Κοινοβουλίου. Αν όμως θέλετε να κάνετε εφικτή τη συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να υπάρξει η υπηρεσία αυτή της εξωτερικής δράσης Οι ανθρώπινοι πόροι θα προέρχονται από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο και από τις ε, αντιπροσωπείες της Κομισιόν στο εξωτερικό. Πρόεδρος, ο κύριος Γκέγερ πάλι δευτερολογεί. Ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου, έχω μια συμπληρωματική ερώτηση Ιδίω πάνω σε αυτό που ερώτησε ο συνάδελφο Ιταλ, έχετε δίκιο ότι τίποτα δεν είναι πιο πολύ πολύπλοκο από την απλούστευση και εισαγωγικά, σαν κατευθύνια γραμμή, αναφερθήκατε στην έννοια ε, του φιλικό και το χρήστη για να μας παρουσιάσετε τις ιδέες σας. Αυτό μου φαίνεται όμως ότι είναι απλώς μια ονομασία. Θα πρέπει να έχουμε ε, σε εθνικές δηλώσεις ε, διαχείρισης από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στον προπλογισμό. Ποια είναι η άποψή σας για τα θέματα αυτά. Grazie. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που συμφωνώ. Θα ήταν καλύτερο για την ευθύνη να έχουμε δηλώσεις των κρατών μελών αλλά είναι και θέμα βούλησης των κρατών μελών. Και χρειαζόμαστε και την πιστοποίηση του εθνικού ελεγκτή. Με διαφοροποίηση από το τι συμβαίνει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Λεβαντόφσκι, η Επιτροπή Ελέγχων του Προπηρισμού έχει σαν στόχο να ελέγχει κατά πόσον πληρωμέ έχουν γίνει σωστά, κατά πόσον υπάρχουν ασθαλίε και είπατε ότι γνωρίζετε το θέμα αυτό πολύ ξεκάθαρα. Τώρα έχουμε ένα νέο κεντρικό θέμα. Δεν θέλουμε να δούμε κατά πόσον πληρωμέ ήταν μόνο σωστέ, αλλά και κατά πόσο ήταν και αποτελεσματικέ. Καλά είναι ο εκ των υστέρων έλεγχο, αλλά δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Θα πρέπει λοιπόν πριν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές θα πρέπει εσεί, παραδείγματος χάρη να εξετάσετε κατά πόσον κάποιο μέτρο μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Τι μπορείτε να κάνετε εσεί για να μπορέσετε να διευκρινίσετε τη θέση σα έναντι των κρατών μελών ιδίω όσον κάποιο μέτρο δεν είναι αποτελεσματικό γιατί πολλά δαπάνε παράλογε πραγματοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Κατόπιν πώ θα συνεννοηθείτε με του συναδέλφου που κάνουν τι μεγάλε δαπάνε, ε, αγροτικά περιφερειακά ταμεία. Έτσι στο παρελθόν φαίνεται ότι δεν ήταν υπαρκή η επικοινωνία με τον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριο Επίτροπο για δύο λεπτά. Το σημείο αφετηρία τη συζήτηση για τι ατασταλίε θα πρέπει να είναι ότι το 2008 η διαδικασία της απαλλαγής έδειξε σημαντική πρόοδο. Είναι πιο δύσκολο εύκολη εισαγωγή του κριτηρίου της αποτελεσματικότητας, γιατί αυτό είναι πιο υποκειμενικό από τα τυπικά κριτήρια. Και είναι πιο εύκολο να γίνει η αξιολόγηση και η κρίση από τυπική άποψη. Κάτι που δεν ισχύει με την αποτελεσματικότητα. Αλλά ο δημοσιονομικός κανονισμός θέλει πια να λάβει υπόψη όχι μόνο μια απλού, απλοποίηση που θα είναι φιλική προς το χρήστη, αλλά και μια ορθολογική απλοποίηση. Τώρα, η ποσοτικοποίηση από, από επιχειρησιακή άποψη είναι πιο δύσκολη. Αλλά, μια και έχουμε τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε και τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις που γίνονται από τα κράτη-μέλη. Γιατί έχουν ξεκινήσει πολλές διαβουλεύσεις, ήδη από πέρυσι τον Οκτώβριο και αν δεν κάνω λάθος έχουν υποβληθεί 200 τροπολογίες για το δημοσιονομικό κανονισμό και πολλές από αυτές προέρχονται από δικαιούχους και ζητούν ε, ακόμη μεγαλύτερη απλοποίηση και όχι συσσόρευση των κριτήριων. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριος Χατζημαρκάκης. Εδώ τα κράτη-μέλη πρέπει να, να δράσουν. Εσείς και στο naming and shaming. ότι ήθεστε να το κάνουν αυτό. Γιατί μόνο αυτό οδήγησε στο μέλλον, όπως είπατε και εσείς, στην βελτίωση και στη μείωση των ατασταλιών. Και ποιο θα είναι το κεντρικό θέμα για σας. Τι είναι πιο αποτελεσματικό για σας, υποδομή ή έρευνα και ανάπτυξη. Κύριε Επίτροπε, έχετε ένα λεπτό. Ξεκινήσαμε ήδη σήμερα την διαδικασία αυτή του name and shame, του ξεμπροστιάσματος των κρατών μελών. Δεν θα ήθελα να γίνει και διμερός. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει και απαριθμίσει ατασταλίες και δεν εκφεύγουν της προσοχής της. Είναι πολύ γνωστά αυτά τα φαινόμενα. Μου θέσετε μία ερώτηση για τις προτεραιότητες προς το ανεκτό περιθώριο λάθους. Η προτεραιότητα είναι η η βελτίωση στις υποδομές, αλλά πολλά παράπονα γίνονται και για την έρευνα, γιατί πολλές αγαθές προθέσεις ακούγονται για την αύξηση των κονδύλων της έρευνας και το 2010 το 1α επλήγει από περικοπή. Μιλούσε για την ανταγωνιστικότητα και αυτό δείχνει, στέλνει ένα πολύ εσφαλμένο μήνυμα για τα ερευνητικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Οι πράσινοι δεν έχουν ε, ορίσει κάποιον ομιλητή. Ο κύριος Τσαρνέτσκι από την ομάδα των μεταρρυθμιστών. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Έκανα λάθος. Η κυρία Τρούπελ θα θέσει την ερώτηση εκ μέρους των πρασίνων για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τώρα μιλούμε για την ε, απλούστευση και πώς θα την ε, βελτιώσουμε ή πώς θα την εφαρμόσουμε. Σας ερωτώ, θέλετε να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη διαχείριση των δημοσιονομικών τους κατά τη χορήγηση των δηλώσεων αξιοπιστίας τους. Για δύο λεπτά ο Επίτροπος. Φοβάμαι ότι πολύ πιο εύκολο θα είναι να συντάξουμε έκθεση Πώ θα βελτιώσουμε εμεί τα πράγματα παρά πώς ε, θα βελτιωθούν οι δηλώσεις αξιοπιστία των κρατών μελών. Στις ερωτήσεις για τις ατασταλίε, ξέχασα να πω ότι διανύουμε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο και έχουμε δύο γύρους απλοποιήσεων, προκαταβολών και την πρόταση για ε, να καταργηθεί η χρηματοδότηση στο κοινωνικό ταμείο, κάτι που δεν δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και διανύουμε και την χρηματοπιστωτική κρίση. Ταυτόχρονα έχουμε τη συζήτηση για το δημοσιονομικό κανονισμό. Η κυρία Γκρέσιλε το ξέρει. Έχουμε όμως δύο γύρους απλουστεύσεων, εφάπαξ ποσών, προκαταβολών. Όλα αυτά τα μέτρα είναι πιο φιλικά προς το χρήστη και δημιουργούν το έδαφος και κάνουν πιο πρόσφορο το έδαφος για την κοινωνική συνοχή, την πολιτική συνοχή και την αντιμετώπιση της κρίσης. Βέβαια δεν ευθυγραμμίζονται πάντοτε με τη χρηστή ε, δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο. Και αυτές οι διαφορετικές ε, τάσεις είναι αντικρουόμενες. Θέλουμε να διευκολύνουμε τα πράγματα τους καιρούς που είναι δύσκολη η πρόσβαση στο δανεισμό από τις τράπεζες. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους δικαιούχους, γιατί αυτό είναι ένα μέτρο για την καταπολέμηση της κρίσης. Απ' την άλλη πλευρά, πιστάμεθα τεράστιες πιέσεις να βελτιώσουμε τη χρηστή μας δημοσιονομική διαχείριση. Μερικές φορές ε, μπλεκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο αλλά θα το αντιμετωπίσουμε σε αυτήν την τριετήρη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Πέραν των νέων μηχανισμών που έχουμε για τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, τα νέα δημοσιονομικά μέσα και την έννοια του ανεκτού περιθωρίου λάθους που θα συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό κανονισμό με συγκεκριμενοποίηση στις διάφορες πολιτικές. Μην ξεχνάτε πάντως ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες λόγω της κρίσης και ψηλέ προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί. Και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις υποσχέσεις μας για τις πολιτικές μέσω της απλοποίησης και των προκαταβολών. Για ένα λεπτό η κυρία Τρούπελ αν θέλει να επανέλθει με συμπληρωματική. Ναι, για το ίδιο πρόβλημα. Συμφωνούμε ότι σίγουρα δεν θέλουμε ε, περισσότερη γραφειοκρατία. Δεν θέλουμε χαρτομάνη αλλά υπάρχει και το θέμα του πολιτικού πνεύματος και της πολιτικής δέσμευσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των ε, δημοσιονομικών. Και πάνω από το 10% υπεύθυνοι γι' αυτό είναι τα κράτη-μέλη. Οπότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, δρα... να δράσουν με κοινό πνεύμα και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την χρηστή διαχείριση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διορθώσουν την δημοσιονομική τους διαχείριση. Και αυτό δεν θα γίνει με αύξηση της γραφειοκρατίας. Το θέμα είναι να αλλάξει η πολιτική παιδεία, το πολιτικό πνεύμα των κρατών μελών, προκειμένου να εφαρμόσουν αυτή τη χρήστη δημοσιονομική διαχείριση. Για ένα λεπτό, κύριο Λεβαντόφσκι. Θα ήθελα να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ανατολική Ευρώπη, όπως λέμε. Ότι δεδομένων των παραπώνων που έχουν διατυπωθεί από την χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, είχαμε τεράστια πείρα με τα προγράμματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κάτι που ήταν καινούριο για τις νέες χώρες. Και βελτίωσε την ποιότητα της ε, διοίκησης στις νέες χώρες. Μπορεί βέβαια να υπήρξαν και πολλές ατασταλίες, όχι κατά ανάγκη στη συνοχή, αλλά εγώ κρατώ την αισιοδοξία μου και προσπαθώ να είμαι θετικός. Πιστεύω ότι υπάρχει βελτίωση σε ό,τι αφορά τη γνώση και το ρόλο των δημοσιονομικών προγραμμάτων, για τον εσωτερικό έλεγχο, για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ακόμη και για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σε πολλές χώρες. Και όχι μόνο για τις παλιές χώρες. Υπάρχει και μία πιο θετική αντίληψη είναι μια επανάσταση αυτή ε, στην ε, τοπική και περιφερειακή διάσταση, στην δική μου περιοχή της Ευρώπης τουλάχιστον, αυτή που γνωρίζω καλύτερα. Μην τα βλέπετε όλα μαύρα. Ο κύριος Σαρνέτσκι από τους μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω σε Πολωνό Επίτροπο φυσικά την ερώτηση στα πολωνικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λεβαντόφσκι για τις καταπληκτικές απαντήσεις που έδωσε στην ε, ακρόασή του και ως συντονιστής της πολιτικής μου, ομάδα, της πολιτικής ομάδας για την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Λεβαντόφσκι που έγινε κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα λάθη σε ό,τι αφορά κάποιες διασπαθήσεις που έγιναν των κοινοτικών κονδύλιων και κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φάνηκαν τέτοια λάθη. Πώς θα διορθώσω αυτή τη διαδικασία, πώς θα την κάνουμε άδεια πέραστη στα λάθη την επόμενη πενταετία. Και δεύτερη σημαντική ερώτηση, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το κόστος της δυνητικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις Βαλκανικές χώρες ό,τι αφορά τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Και σας εύχομαι και καλή επιτυχία κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο Επίτροπος έχει το λόγο. Νομίζω ότι αυτό είναι ε, υποδειγματική περίπτωση ε, δύο ανθρώπων που στην εθνική πολιτική είναι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά με, ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη αυρότητα συζητούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα υπάρχουν κάποια λάθη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των προϋπολογισμών. Και υπάρχουν δύο τομείς όπου δυστυχώς η εφαρμογή είναι λατωματική, προβληματική. Ο πρώτος τομέας είναι η συνοχή. Αναφέρθηκε ότι εκεί υπάρχει το υψηλότερο επίπεδο τασταλιών. Το δεύτερο είναι οι εξωτερικές ε, δράσεις. Ε, αυτοί οι δύο τομείς παρουσιάζουν τα περισσότερα λάθη και εκείνη που θα πρέπει να βελτιώσουμε τον ορθολογισμό της δημοσιονομικής διαχείρισης και διασπάθηση και σπατάλη συνήθως κάνει μια διοίκηση που έχει μικρή συμμετοχή στον κοινοτικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά όχι μόνο τον έλεγχο των λογαριασμών αλλά και κάποιους τομείς που αφορούν άλλες κατηγορίες και ενώ σε ορισμένες ε, τομείς υπάρχουν πολλές ατασταλείς, σε άλλες ε, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διεύρυνση και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό που μας τραβά την προσοχή είναι κυρίως ότι υπάρχουν κάποια επίμαχα προβλήματα με την ένταξη της Τουρκίας που αν ενταχθεί θα απορροφήσει το 60% των διορθωτικών κονδυλίων σε σχέση με όλες τις χώρες που βρίσκονται σε τροχιά ενταξιακής ή προενταξιακής διαδικασίας. Επίσης ε, δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις για το κόστος ένταξης της Τουρκίας. Δεν θα ήθελα να σας ε, προβληματίσω με τους αριθμού αυτούς, γιατί ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να γίνει πρόβλημα για τον προϋπολογισμό του 2010. Δευτερολογία κύριο κύριος Τσαρνέτσκι. Σας ευχαριστώ για την ε, ενδιαφέρουσα απάντησή σας. Ε, σίγουρα οι δαπάνες της διοίκησης είναι α, ε, αντίστοιχες με τις εξωτερικές ε, δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αλλάξει όμως αυτή η αναλογία. Και αυτό είναι και δικό σας έργο. Γι' αυτό και σας εύχομαι καλή επιτυχία, παραλαμβάνω κύριε Επίτροπε, και ευελπιστώ ότι θα είναι πολύ αποτελεσματικό το έργο σας στην επόμενη Επιτροπή. Ο Επίτροπος. Όντως, σίγουρα η κατηγορία 5 είναι λίγο ανώτερη στον όγκο της από την κατηγορία 4. Το, η κατηγορία 4, το κεφάλαιο 4 αυτή τη στιγμή είναι προνόμιο και της ε, Επιτρόπου που θα υποστεί ακρόαση παρόμοια με εμένα, της κυρίας Άστον. Και μιλούμε για ένα κονδύλιο 45 δις ευρώ. Βέβαια ακόμη δεν έχει ε, επιληθεί το θέμα της οργάνωσης ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της ΓΚΟΕ, το λόγο κύριο Σόντεγκορτ. Ή απουσιάζει. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ για να θέσει ερώτηση. Ο κύριος Πόρτες. Εδώ Μιλούμε για την αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη διόρθωση, τη μείωση των ατασταλιών και τον περιορισμό της πατάλης. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας αποτελεσματικότητας που αφορά την επιλογή, ε, τις πολιτικές μας επιλογές και τις συνέπειές τους ε, στον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, πολλές ε, κατηγορίες του προϋπολογισμού οφείλονται σε πολιτικές συμφωνίες που γίνονται μεταξύ διαφόρων συμφερόντων. Ερωτώ λοιπόν, Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να συζητηθεί αυτό που λέμε δημοσιονομικές προοπτικές μηδενικής βάσης για να γίνει μια ανακατανομή των προτεραιοτήτων και των ε, μηχανισμών και εργαλείων της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο Επίτροπος. Τώρα, για το μέλλον και τις μελλοντικέ δημοσιονομικές προοπτικές. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και το δίδαγμα του παρελθόντος, που μας λέει ότι όσο πιο νωρίς συγκεκριμενοποιήσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες, το πιο εύκολο θα είναι να τις εφοδιάσουμε και με δημοσιονομικά μέσα. Βέβαια το πρόβλημα είναι πώς θα βρούμε τον κεντρικό μας προσανατολισμό. Θα μπορούσε να είναι οι κλιματικές συνθήκες, για παράδειγμα, το περιβάλλον αλλά θα πρέπει να έχει απήχηση αυτή η προτεραιότητα και στο κοινό. Και τα προηγούμενα πακέτα είχαν, είχαν κεντρικούς προσανατολισμούς, για παράδειγμα την εσωτερική αγορά. Το πρώτο πακέτο Delors, μετά η νομισματική ένωση για το δεύτερο πακέτο Delors. Κατόπιν είχαμε την Επιτροπή Πρώτη που είχε ως προτεραιότητα και κεντρικό προσανατολισμό τη διεύρυνση με ανάμεικτα ανάμικτα συναισθήματα στην Ευρώπη. Τώρα η πρώτη Επιτροπή Μπαρόζο επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα τη Λισαβόνα. Δεν προκάλεσε όμω και πάρα πολλά θετικά συναισθήματα. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα με το ποιο θα είναι ο κεντρικό προσανατολισμό τη δεύτερη επιτροπή Μπαρόζο. Και πού θα πρέπει να επικεντρώσουμε τι πολιτικέ μα προτεραιότητε και τις ε, προτεραιότητες των δημοσιονομικών μας προοπτικών. Αυτό θα το καλύψουμε και με την αναθεώρηση. Αλλά η αναθεώρηση καθυστερεί. Και αυτή ήταν πολύ σοφή η απόφαση να εκχωρηθεί η αναθεώρηση, να μεταβιβαστεί στην επόμενη Επιτροπή. Δεδομένου όμως ότι ο κύριος Μπαρόζο θέλει να εγκριθεί πρώτα η στρατηγική για το 2020 και αυτή είναι η πολιτική προτεραιότητα, και αυτό θα γίνει μάλλον τον Ιούνιο, κατά πάσα πιθανότητα το νωρίτερο η αναθεώρηση αρχίσει τον Ιούλιο. Αν συνδυαστεί και με την ταξινόμηση των προτεραιοτήτων από πολιτική άποψη. Οπότε πλησιάζουμε ήδη στο χρονοδιάγραμμα της επόμενης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και το θέμα της παράτασής του. Αλλά αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Πόρτας για ένα λεπτό. Ναι. Δράτω με τις ευκαιρίες που μου δίνει με την απάντησή του ο κύριος Επίτροπος. Ακριβώς επειδή πλησιάζουμε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία της αναθεώρησης αυτών των δημοσιονομικών προοπτικών, διευρύνοντας χρονικά μέχρι το 2015-2016 και να έχουμε γνήσιες πραγματικές νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Πρέγκο, Παρακαλώ, ένα λεπτό. Φοβούμαι ότι η ερώτησή σας είναι η ερώτηση κάποιου που ε, θέλει απλή παράταση. Και αυτό θα επαναλάβω. Μία από τις λύσεις του προβλήματος του συνολισμού της ε, εντολής του Κοινοβουλίου με τις δημοσιονομικές ε, θα ήταν καλό. Η ιδέα μου να παρατηθεί η θητεία του Κοινοβουλίου σε 7 χρόνια δεν έγινε αποτεκτή. Αν θέλετε εσείς τώρα συντονισμό ε, σε αυτή την ετή περίοδο αυτό στη συνθήκη λέει τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ίσως μία παράταση είναι δυνατόν να συζητηθεί. Αλλά δεν είναι η μόνη δυνατότητα για το συντονισμό των δύο. Είναι όμως μία από τις ε, προτάσεις. ευχαριστώ. Ο κ. Ανδρεάσεν είναι παρόν και δεν είναι παρόν άλλον και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φερνάρο. Α, αν απουσιάζει τελειώσαμε κύριε Πρόεδρε. Merci, Monsieur le Président. Je suis très... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντυπωσιάζομαι τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα της, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του και ο Πρόεδρος τους σέφονται τους κανόνες. Είμαι πεπισμένος ότι τώρα τα μέλη της Επιτροπής Προπολισμών θα φροντίσουν να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο εξ ονόματος του ΕΛΚ στον κύριο Ράιμε Μπέγκε. Ο κύριος και ξέρει ότι γεωγραφικά είναι κατά κάποιον τρόπο ανάμεσα στους δύο διαδόχους του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε γνωρίσαμε τον προεδρόμενο επίτροπο σαν πρόεδρο τη Επιτροπή μα, αλλά και σαν επικεφαλή των διαπραγματεύσεων των δημοσιονομικών προβλέψεων. Γι' αυτό εκ των προτέρων λέω ότι η ικανότητα τη εξουσία και η κοινοβουλευτική του ανοιχτή στάση δεν αμφισβητούνται. Παρόλο αυτό γνωρίσαμε και δύο ότι σε δύσκολε στιγμές των διαπραγματεύσεων αυτών το 2006 το σύνολο της Επιτροπής δεν κάλυψε επαρκώς τις δικές της προτάσεις. Και γι' αυτό έχουμε ελλείμματα και κατάλοιπα τα οποία συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον κύριο Λεβαντόση καταρχήν όσον αφορά την εφαρμογή των δημοσιομικών επιπτώσεων από τη θήκη Λισαβόνα. Πότε οι υπηρεσίε θα αξιολογήσουν περίπου τους πόρου που θα χρειαστούμε για την εφαρμογή του Λισαβόνα, όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική, αλλά και για όλε τι νέε πολιτικέ προτεραιότητες. Και δεύτερον, η προβλεπόμενη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση δεν θα μπορούσε να εξτάσει το θέμα της παράτεσης και επανεξέτασης των πολιτών προγραμμάτων και μεγαλύτερης ευελιξίας στα μέσα δεν θα πρέπει να εξεταστεί τώρα αυτό το θέμα και όχι μετά το 2014. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λεβαντόφσκι, ένα λεπτό. Ο, δύο λεπτά, συγγνώμη. Ο Ράμερ Μπέγκερ με βοήθησε όταν μάθαινα επί τόπου τι πρέπει να κάνω το 2004. Όσον αφορά τις προσαρμογές της ενδείξης αγώνας, το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό. Σύντομα όμως θα είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε εκτός από τις μεταφο... προσωρινές ε, προτάσεις για μεταφορά πόρων και ρεαλιστική διαδικασία που συμφωνήθηκαν στην Λόγω Επιτροπή, περιμένοντας όμως τη μεταφορά του πρωτογενού δικαίου σε νόμιμα δεσμευτικές διατάξεις για τις δημοσιονομικές προβλέψεις και μια διαθεσμική συμφωνία. Θεωρώ ότι αυτά δύο έγγραφα είναι πολύ σημαντικά. Συζητούνται τελικό στην Κομισιόν, χρειάζονται και τα δύο. και το Συμβούλιο μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου ε, εξετάζει το θέμα των πολιετών πλαισίων και τον κανονισμό. Η διαθεσμική συμφωνία θα πρέπει να είναι η ευκαιρία και η έκθεση για την διαθεσμική συμφωνία θα είναι η ευκαιρία το τι μπορούμε να κάνουμε με συμπληρωματική ευελιξία. Μέσα δηλαδή το μέσο έκτακτης ανάγκης, ε, αλληλεγγύης και ούτω καθεξής. Ε, όλα αυτά μέσα στα πλαίσια πολύ στενών περιθωρίων όμως των σημερινών προβλέψεων. χτάχτη σας το είπα εισαγωγικά, αλλά εγώ θα ήθελα τα ανώτατα επίπεδα να ξεπεράσουν αυτό το περιθώριο. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε συμπληρωματικές ανάγκες. Έχουμε τρεις φορές αναθεωρήσει τις δημοσιονομικές προβλέψεις. Το 2006 έγινε κάτι που εγώ θα ήθελα να το ξεχάσω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ράιμερ, όχι, δεν θέλει να δευτερολογήσει. Αντιπρόεδρο, κυρία Γιούτα Χάουκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Συχνά ε, ασχολούμαι με το θέμα των εξωτερικών υπηρεσιών και τώρα ξέρουμε ότι οι υπηρεσίε αυτέ δεν μα έρχονται ελονοκοτεύοντες τις δημιουργούμε εμείς. Εσείς, κύριε υποψήφια επίτροπε, πώς εκτιμάτε τη σημερινή κατάσταση. Όπως ορισμένοι από τους συναδέλφους σας ή και τους συναδέλφους μου θεωρείτε ότι ανεξάρτητα αυτές οι υπηρεσίες είναι ένα τμήμα της ε, κοινοτικής ε, διοίκησης και αποδυναμώνουν την εφαρμογή της ε, κοινοτικής πολιτικής. Εάν ναι, θέλετε να το αλλάξετε και πώς θα το αλλάξετε. Αν όχι, φαντάζομαι θα θεωρείται πολύ σημαντικό, όπως και εγώ, να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διοίκηση, όχι μόνο των υπηρεσιών, αλλά του συνόλου της Κομισιόν και των υπηρεσιών της Κομισιόν. Και εάν δεν συμφωνείτε, θεωρείτε ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα πρέπει να εξετάσει το θέμα της χρηματοδότησης των νέων υπηρεσιών, όχι μόνο το νομικό πλαίσιο και ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει μια κατηγορία ή υποκατηγορία για όλες αυτές τις υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια της νέας απόφασης. Ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ. Δύο λεπτά και Λεβαντόφσκι. Η ανάπτυξη αποφασης ευχαριστω σε ευχαριστω δυο λεπτα και λεβαντοφσκι η αναπτυξη αυτων των δεκανοστικών υπηρεσιών ήταν μια εξέλιξη ad hoc Μετά το 2004 όμως με τη δικιά σας συμμετοχή έχουμε τακτικά την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Όσον αφορά την δημοσιομική διάσταση στο μέλλον, δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από την εφαρμογή στον πληθωρισμό και του πραγματικού κόστους εκτός από το θέμα της Λαροζιέρκ 2 στα 40 εκατομμύρια νομίζω που είναι συμπληρωματικό κόστος για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες για την ε, επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, πράγμα που είναι η επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όσον αφορά τη διαχείριση, πολλά ξέρουμε. Ποιοι είναι οι παράμετροι που λείπουν που παράμετροι που προσανατολίζονται στη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών και υπήρχε μια σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν από το περασμένο έτος. Η διαθεσμική ομάδα καθορίστηκε η κυρία Χάουκ είναι στην υπηρεσία αυτή, η Γκάμπου Γκέσλε είναι, αν είναι εκεί, συναντούν σε επίπεδο αυτής της διαθεσμικής ε, ομάδας για να βελτιώσουν τις ελλείψεις αυτές της διαχείρισης. Αλλά ένα από τα συμπεράσματα και είναι κάτι που προέρχεται από το κοινοβούλιο ίσως αλλά ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ο ευρωπαϊκός προπολισμός να είναι πιο ευέλικτος είναι να έχουμε λιγότερους τίτλους για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Μια ιδέα μου είναι και αυτό. Για να μην υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολύ υπότιτλοι στον προπερισμό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Άλβαρο, Αντιπρόεδρος. Uh, Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ο πρόεδρος Μπαρόζο μεταξύ άλλων κυρίων προτεραιότητων αναφέρθηκε στο εξή. Το ένα είναι η οικονομική και ε, δημοσιονομική κρίση και το άλλο είναι τα προβλήματα που ανεπιτρέπουμε εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών. Όσον αφορά την χρηματοπιστική κρίση, θα ήθελα να έχω τι δικέ σα απόψει όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Θεωρείτε ότι είναι επιτυχέ ο μηχανισμό για τη χρηματοδότηση για το συγχρηματοδότηση μάλλον έχει επιλεχθεί σωστά και κατά πόσο θα καταλήξει σε μια γραμμή του υπεροπλογισμού στο μέλλον, αν το θέλουμε αυτό, ή θα έχουμε άλλη νομική βάση. Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν. Το άλλο θέμα είναι η έρευνα και η ανάπτυξη και θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το χρονικό πλαίσιο και η προσωρινή εξολόγηση του ερευνητικού πλαισίου του 2007 Πώς θα μπορούσε καλύτερα να δούμε κατά πόσον ωφελούμεθα από τα χρήματα αυτά της έρευνας. Ποιες είναι οι δικές σας προσωπικές ιδέες επίσης για το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 8. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κ. Λεβαντός για να απαντήσει. Το Ταμείο Αποκοσμιοποίησης ε, καθεντρήθηκε ίσως για να αποκριθεί σε ανησυχίες που εκφράστηκαν στα πλαίσια του γαλλικού δημοψηφίσματος. Αλλά τώρα όσο πάει και περισσότερο χρειάζεται, παραδείγματος χάνει το θέμα και της απασχόλησης. Και συζητάμε πραγματικά το θέμα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης όσον αφορά τους κανόνες για κάποιους περιπτώσεις Θυμάστε την περίπτωση της ΣΤΕΛ που ήθελε να μεταφερθεί από την Ιρλανδία και το θέμα της ε, δημόσιας για το Ντουβάντσο στη χώρα μου στην Πολωνία. Αυτό που χρειάζεται είναι κάποια τροποποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης για να μην υπάρχουν επικαλύψεις όσον αφορά τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων ή αιτήσεων για χρηματοδότηση από το αυτό, αλλά να υπάρχει ένα διαφορετικό σύστημα για να μπορεί κανένας να έχει πρόδοση στα χρήματα αυτά. Αυτό είναι θέμα βέβαια και στη διακριτική ευχέρεια και όποιος έρθει πρώτος είναι εκείνος που παίρνει πρώτος τα χρήματα. Στο Γκτάνσκ, στη πόλη μου, κατασκευάζεται ε, μια εγκατάσταση που δεν μπόρεσε να φτάσει <clears throat> να ζητήσει χρήματα από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, πράγμα που ήταν σφάλμα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε στις μελλοντικές δημοσιονομικές προβλέψεις τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή. και θα πρέπει αυτό να αναφέρεται στην αναθεωρημένη δια... θεσμική ε, ε, συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να απαντήσω στη συμπληρωματική σας ερώτηση. Πρόεδρος, εάν ο στόχος του Τομείου Παγκοσμιοποίησης ήταν να είναι δημοφιλή, η παγκοσμιοποίηση στη Γαλλία, απέτυχε πλήρω. Ο κύριος Αλβάρο μπορεί να δευτερολογήσει. Ναι, ευχαριστώ. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε όλοι ζητάνε χρήματα από το Ταμείο Αποκοσμιοποίησης, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Κατά πόσον αυτό έρχεται σε αντίθεση ή δεν έρχεται σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ξέρετε τις διαδικασίες. Ε, και επίσης ε, μπορείτε τώρα να αναφερθείτε στο θέμα της ε, έρευνας και της ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Βαντόφσκη θα απαντήσω, στο θέμα της έρευνας και ανάπτυξης. Εξετάσαμε λίγο για το θέμα της ε, διαθεσιμότητας. Εδώ έχουμε πολλές σημαντικές δηλώσεις για το μελλοντικό προεπλογισμό. Είτε θα μπορούσε σαν πλαίσιο χρηματοδότησης να είναι περισσότερο από εκείνο που μπορούμε εμείς να υπομισθούμε. Και Επίσης, έχουμε και μικρότερα προβλήματα στον τομέα της έρευνας. Yes, um, I would like um, to... Θα επανέλθω σε μερικές ομιλίες στο Κοινοβούλιο πρόσφατα κύριε Λεβαντόφσκι όπου είπατε ότι το περιβάλλον είναι σε... κάνει ζημιά στην οικονομική ανάκαμψη. Και αυτό μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στις νέες γραμμές στον προπολογισμό. Έχουμε απόδειξη ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ότι είμαστε, αν είμαστε έξυπνοι και συνδυάσουμε την βιωσιμότητα, την πράσινες τεχνολογίες, θα έχουμε νέα απασχόληση, νέα οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη. Είστε διατεθειμένος να αλλάξετε την άποψή σας. Ο κύριος Λεβαντόφσκι, δύο λεπτά. Σας συγχαίρω για την προετοιμασία σας. Έχετε ήδη τρία καπέλα που φορέσατε στην σημερινή ακρόση. Όντως, εγώ αναφερόμενα στο πρόγραμμα σε μια χώρα η οποία στηρίζεται στη χρήση του άνθρακα. Η χώρα μου, η χώρα μου είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Η Πολωνία είναι χώρα που πιστεύει στην Ευρώπη, αλλά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει σχέση με την ε, θέρμανση του πλανήτη. Πάνω από το 90% των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού στηρίζεται στη χρήση άνθρακα. Σωστά είπατε ότι η ευκαιρία αυτή εν μέρη συγχρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα ανάκαμψης για νέες τεχνικές εναποθήκευσης, εξαέρωσης και συμφωνώ και στο σημείο αυτό αλλάζει ενδεχομένω η θέση μου, συμφωνώ ότι η πράσινη βιομηχανία είναι μια από τις πιο πολλά υπεσχόμενες βιομηχανίες στην Ευρώπη και στηρίζεται σε επιχειρήματα υπέρ του περιβάλλοντος. Αυτό το κατανοώ, διότι τώρα βλέπω και στην Πολωνία τη σοβαρή προσπάθεια να, κρατήσουμε, να είμαστε στο ύψος των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Παρά το ότι ο άνθρακας είναι μια, ένας φυσικός πλουτοπαραγωγικός πλούτος, ε, πόρος της χώρας μας. Αλλά η τεχνολογία οι νέε τεχνολογίε επιτρέπουν, παραδείγματο χάρη, πιλωτικά προγράμματα εξαέρωση κλπ. που είναι τμήμα του, προγράμμα, του προγράμματο οικονομική ανάκαμψη. Είναι μια ευκαιρία αυτό. Είναι όντω μια ευκαιρία για την Πολωνία. Πρόεδρο. Στην εκλογική μου περιφέρεια αυτή τη στιγμή εγκαινιάζεται το, το πιλωτικό πρόγραμμα σύλληψης και αποθήκευσης του άνθρακα και η ακρόση σήμερα με εμπόδισε να είμαι παρόν στην ιστορική αυτή στιγμή στη χώρα μου. Η κυρία Ντουιρόν. Κύριε υποψήφε επίτροπε, είπατε ότι ασχοληθήκατε με τις μεταρρυθμίσεις για τα λιμάνια στην Πολωνία και διάβασα και τις δηλώσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα. Τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους απελευθερωμένους τομείς και τις κρατικές ενισχύσεις την κρατική ρύθμιση και τη θέση της Ένωσης ως προς αυτό. Ποια είναι η θέση Δηλαδή, από μια μεριά έχουμε τον ανταγωνισμό που έχει σχέση με την αναδιάρθρωση τομέων και από την άλλη το όραμά σας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και πώς μπορεί να τις πλαισιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση ενός λεπτού. Το πιο καλό εργαστήρι γι' αυτό είναι η Πολωνία η οποία πλήγει όσον αφορά την, τα μεγάλα ναυπηγεία με έντονο ανταγωνισμό μάλλον με τον, με τον νόμο περί ανταγωνισμού της Ένωσης. Συμφωνήσαμε με τη λογική του, της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό. Δεν μπορείτε να στηρίξετε την ανταγωνιστική, τας, σας θέση με κρατικά κονδύλια. Αυτό δεν γίνεται. Είναι στρέβλος το ανταγωνισμό αυτό. Δεν είναι πραγματικός ανταγωνισμός. Ωστόσο, κατανοώ και κατανόηση κατά κάποιο τρόπο είναι ένα είδος Δηλαδή είναι δύσκολο να περάσουμε από τη μία μέρα στην άλλη από τις ρυθμίσεις που υπάρχουν, που υπήρχαν μάλλον, στις νέες. Η αλλαγή πρέπει να γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό μιλάει για εργαστήρι όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Τρία μεγάλα ναυπηγεία στην Πολωνία έχουν κλείσει, σας θυμίζω. Ο κύριος Πάβες Κόβαλ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχετε το λόγο κύριε Κόβαλ. Δύο, όχι ένα. <coughs> Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της χρηματοδότησης της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Ποια είναι η θέση σας. Τι χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να αφιερωθούν στην εξωτερική πολιτική που θα είναι και το νέο τέκνο της, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Αναφερθήκατε και στο θέμα της χρηματοδότησης της ανατολικής εταιρική σχέσης, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Δυστυχώς είναι τα κονδύλια που αφιερώνονται σε αυτό, ιδιαίτερα αν δούμε την ε, κατανομή τους ετησίως. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης σας για το θέμα αυτό και ποιο είναι το βέλτιστο επίπεδο χρηματοδότησης των σχεδίων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ώστε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικός παίκτη σε ό,τι αφορά τη δέσμευσή μας ε, και να είμαστε ανταγωνιστικό παίκτη σε σχέση με την Ρωσία που έχει ενδιαφέρον και αυτή στην περιοχή. Σα ευχαριστώ κύριο Λεβαντόφσκι για δύο λεπτά. Το θέμα, η κατηγορία 4, η εξωτερική πολιτική, το κεφάλαιο 4, είναι το πιο χαρακτηριστικός πονοκέφαλος, η μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά των ετήσιων διαπραγματεύσεων και της αναθεώρησης και των πολύ σφοδρών συζητήσεων για τον προπολογισμό. Γιατί κάθε φορά έχουμε όλο και περισσότερε ε, αποστολέ και καθήκοντα που δεν εντάσσονται στα ανώτατα όρια των δημοσιονομικών προοπτικών. Και δεν έχουμε μόνο την Ανατολική Εταιρική Σχέση, έχουμε και το Κωσυφοπαίδιο, έχουμε την Παλαιστίνη, έχουμε και άλλες ε, απροσδόκητες ανάγκες ή ευνίδιες ανάγκες που ανακύπτουν και ζητούν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό. Σε ό,τι αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, ήταν στην αρχή μία από τις πολιτικές που αναγγέλθηκαν ως ε, αρχή, ε, αλλά δεν είχαν ε, πρικοδοτηθεί με χρηματοοικονομικά μέσα. Τώρα έχουμε κάποια κονδύλια για την πολιτική της γειτονίας και έχουμε 600 εκατομμύρια ευρώ για την πολιτική της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αυτά τα κονδύλια δεν προέρχονται από νέα ε, από νέες πηγές. Δεν είναι νέα χρήματα, δεν είναι φρέσκα χρήματα. Είναι, ανα, είναι αναδίπλωση, είναι περιθώρια. Δεν βρέθηκαν καινούρια κονδύλια. Έγινε ανακατονομή των κονδύλιων. Τα 600 εκατομμύρια είναι μικρό ποσό και η γεωγραφική επικράτεια είναι τεράστια. Αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις, ε, τα κονδύλια αυτά πρέπει να βρούμε ε, κονδύλια εκτός του κοινοτικού προπολογισμού. Το 2010 και ίσω και το 2011 δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Γιατί δεν υπάρχουν πια περιθώρια ελιγμών και διακριτική ευχέρεια σε αυτή την κατηγορία 4. Και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αισθητή αύξηση των κονδύλιων για την ανατολική εταιρική σχέση. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοποίηση των κονδύλιων, σε ό,τι αφορά του δικαιούχου, τότε εσεί κύριε Κόβαλ νομίζω ότι για το θέμα αυτό έχετε πολύ πιο ειδικέ γνώσει. Θέλετε συμπληρωματική ερώτηση κύριε Κόβαλ. Όχι, σας ευχαριστώ. Η κυρία Μιχαήλοβα Νιέμσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαντόφσκι. Ο κύριος Λόζεβιτς ήδη εξάντλησε την ερώτηση που θα είχα να σας κάνω. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας κάνω κάποια ερώτηση. Είπατε ότι η Κομισιόν θα αναθεωρήσει επιγόντως το δημοσιονομικό κανονισμό με βάση την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία Μπορείτε να μας πείτε τουλάχιστον ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα περί αυτού. Και δεύτερο, το ρόλο σας ως Επιτρόπου στο διάλογο με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε θέματα κοινή εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Πώς τον βλέπετε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δύο λεπτά ο κύριος Λεβαντόφσκι. Δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Δεν είναι εύκολο για το δημοσιονομικό κανονισμό και την αναθεώρησή του. Και θα γίνει πολύ γρήγορη, ταχεία αναθεώρηση με βάση και το πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τον προπολισμό του 2010 ζητεί όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την οικονομική αναθεώρηση να γίνουν σε βάση τριετή Αλλά αυτό δεν αναφερόταν σε αυτό που λέμε fast track revision, ταχεία αναθεώρηση. Αν θέλουμε γρήγορα να συσταθεί αυτή η υπηρεσία μέχρι τέλος Απριλίου, όπως σας είπα πριν, θα πρέπει να έχουμε υπερταχή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Αντίθετα με αυτό που θεωρεί η Ίνγκε Γκρέσλε, γιατί γνωρίζω τη θέση της. Το πραγματικό πρόβλημα σας το είπα. Θα πρόκειται για ένα ανεξάρτητο όργανο σε σχέση με το δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι υπεύθυνο για τις διοικητικές του δαπάνες. Αλλά οι λειτουργικές δαπάνες και επειδή απάντησα ήδη εν μέρη σε αυτό, πάντως με βάση την λογική της πλήρους ευθύνης της Κομισιόν για τις λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει να ελέγχεται και να είναι τμήμα του προπολογισμού της Επιτροπής. Το πιο σημαντικό και στις δύο αυτές τις τα δύο σκέλια αυτά, το διοικητικό σκέλος και το λειτουργικό σκέλος, θα είναι πλήρως υπόλογο έναντι του Ευρωκοινοβουλίου όσον αφορά την απαλλαγή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλφίν, Αντιπρόεδρος, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λιμανταυσκή, όλοι ξέρουμε ότι οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης δεν επαρκούν όσον αφορά τον προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση σήμερα και αύριο, γιατί συνεχίζεται. Πρέπει να μεγιστοποιηθεί λοιπόν η χρήση αυτών των πόρων και μια πιθανή λύση θα ήταν να αυξηθεί η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή. Ο κ. Μπρόσο ζήτησε μεγαλύτερο μείγμα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ταμείων και των δανείων αυτής της τράπεζας. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και ρωτώ ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης ο κύριος Μπαρόσο δεν είναι υπερβολικά φιλόδοξος όσον αφορά τους στόχους αυτούς για την Ένωση. Όσον αφορά την έρευνα, βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 2010, τι προβλέπετε και θα μπορούσε να υπάρχουν νέα μέσα για να διευκολυθεί η πρόσβαση στα κοινωτικά κονδύλια και μακροπρόθεσμες επενδύσεις παρά την έκκληση του κύριου Μπαρόσο περί του αντιθέτου. Πρόεδρος. Ο κύριος Νεβαντόφης θα μας απαντήσει σε δύο λεπτά. Το κύριο όχημα για απάντηση του κοινωτικού προπολογισμού στην οικονομική κρίση είναι το πρόγραμμα ανάκαμψης, recovery plan. Καθυστέρησε κάπως 5 δις ευρώ σε σχέση με το τονοτικό πακέτο των εθνικών κυβερνήσεων Δηλαδή, παράλληλα πέραν της ερώτησής σας, θα πρέπει να αναφέρουμε και την, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που υπάρχουν. Πάμε χάρη η απόφαση να δοθούν προκαταβολικά πάνω από έξι δις για τη συνοχή. Ήταν ένα, ένα μέσο για να καταπολεμηθεί η κρίση. Τώρα, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο ρόλος της αυξάνει. Σκόπιμα να αυξηθεί η κεφαλαιοποίησή της, να αυξηθεί η δυνατότητά της για δράση και να δοθούν επιστώσεις παραδείγματο χάρη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει νομική υποχρέωση του τραπεζικού συστήματος που ωφελείται από τα δάνεια της τράπεζας να δώσουν διπλάσιο ποσό από αυτό που παίρνουν ως δάνειο. Αυτό είναι μια υποχρέωση συμβατική των τραπεζών. Αυτό ήταν ένας τρόπος. Οι πιστώσεις 75 δις ετησίως μόλι τη δράση μόχλευσης που έχει, δηλαδή έχουμε δύο, 200 δις ευρώ λόγω της μόχλευσης αυτής, Άρα συμφωνώ να υπάρξει αυτή η δυνατότητα ε, περαιτέρω αυξημένης δράσης του κοινωνικού προπολογισμού. Πρόεδρος. Ο πρόεδρος Μπαρόσο από ό,τι πληροφορούμε, επιφόρτησε τον κύριο Καμτεσί, πρώην Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με αποστολή να μελετήσει και να προτείνει το πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να συμβάλλει κι άλλο στη χρηματοδότηση εκτός Ένωσης. δευτερολογία του βουλευτή. Αν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενισχυθεί, θα προτείνετε κάποια μέτρα για να μην επιτρέπει παράλληλος προϋπολογισμός στην, στον κοινωτικό προϋπολογισμό, γιατί αν έχουμε σε παράλληλα μέσα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ακόμη και στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα, τότε η δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης ίσως ε, διακινδυνεύσει να έχει και ένα παράλληλο προπολογισμό, κάτι που είναι εις βάρος της διαφάνειας. Δεν νομίζω ότι με τέτοια μέσα θα προωθούν οι πολιτικές της ε, κοινότητας. Ο κ. Λεβαντόφσκι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα διεθνές νομισματικό ταμείο για τη ζώνη ευρώ. Κάτι που αναβαθμίζει κατά πολύ το ρόλο της ΕΤΕ. Πάντως, αν θέλει η να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να, να λάβει υπόψη κάποια κονδύλια από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Τώρα, μια και πρόκειται για δημόσια κονδύλια, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Είναι θέμα ελέγχου των, ε, κρατικό, των δημόσιων δαπανών. Και σε πολλές χώρες, ακόμη και στην πατρίδα μου, έχουμε προβλήματα η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ε, Πολωνία δεν λειτουργεί γιατί υπάρχει μια προκατάληψη με την ανάμειξη του ιδιωτικού φορέα. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπήρξαν προβλήματα και με απάτες. Γι' αυτό και είναι δύσκολο για μια χώρα που τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθεί να δημορφώσει μια νέα μορφή το, της δημόσιας διοίκησής της. Αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο. Αν θέλουμε να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας, ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι τα νέα δημοσιονομικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός και φορέας. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην ερώτηση του κυρίου Γκοντμάνης. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πώς θα ολοκληρώσουμε τις προηγούμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, στο Κοινωνικό Ταμείο και το Αναπτυξιακό Ταμείο για την περίοδο 2000-2006, γιατί τα 4,45 δισεκατομμύρια ευρώ δεν θα προλάβουν να απορροφηθούν από τα κράτη-μέλη. Και έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό απορρόφηση. Το Ταμείο Συνοχής θα ολοκληρωθεί φέτος και ίσως περισσέψουν 16 δισεκατομμύρια. Οπότε το 4,45 το περίσσευμα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Κάτι που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, τήρησαν τις υποχρεώσεις τους από τις δημοσιονομικές προοπτικές. Πώς θα χρησιμοποιηθούν λοιπόν αυτά τα κονδύλια. Θα χρηματοδοτήσουν άλλες ανάγκες, την παγκοσμιοποίηση για παράδειγμα ή άλλη προτεραιότητα. Ή θα επιστραφούν στα κράτη-μέλη. Δεν είναι σαφές τι θα γίνει με τα κονδύλια αυτά. Ποια είναι η γνώμη σας. Πολύ σαφής ερώτηση. Έχετε δύο λεπτά κύριε Λεβαντόφσκι. οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις και η μη απορρόφησή τους είναι απόδειξη ότι δεν τηρήθηκαν αυτές οι υποχρεώσεις και απόδειξη ότι δεν υλοποιήσαμε τους στόχους μας σε ό,τι αφορά αυτές τις πολιτικές. Το μείζον πρόβλημα ή μάλλον αυτά τα ράλ που μένουν, τα υπόλοιπα για τις εκρεμείς αναλήψεις ε, υποχρεώσεων εμπίπτω στη λογική του νήσιν 2, νήσιν 3 για ορισμένε χώρε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αναλάβω δέσμευση. Και είναι γνωστό το πρόβλημα. Τι θα γίνει με την ανακύκλωση των κονδυλίων, κάτι που είναι πολύ δύσκολο δεδομένη της κρίσης και των δημοσιονομικών ελλημάτων στις, ε, στη ζώνη των ε, καθαρών πληρωτών ή το decommitting, η απομάκρυση από τις αναλήψεις. Έχουμε το σημείο 17 της ε, διοργανικής συμφωνίας για την αναβάθμιση κάποιων κονδυλίων και ποσών, ιδιαίτερα για ορισμένε χώρε όπως η πατρίδα μου. Πάντως, μην περιμένετε από μένα τώρα απάντηση, είναι θέμα συλλογική ευθύνη του Σώματος των επιτρόπων. Εγώ θα προσπαθήσω πάντως να επιλύσω αυτό το πρόβλημα που το απαριθμίσατε σαφέστατα και είναι και ποσοτικοποιημένο. Ο κύριος Γκοντμάνης, για ένα λεπτό. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε κατά 10% ε, στο Ταμείο Συνοχής και στο Αναπτυξιακό Ταμείο τις προκαταβολές για να αντιμετωπίσει την ε, ύφεση. Υπάρχει όμω ίσω πρόβλημα με την Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχων Προπολογισμού. Και εξαιτία τη ε, χαμηλή πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό ζητήθηκε ε, μείωση του ποσοστού συγχρηματοδότηση των κρατών μελών. Οπότε θα υπάρξει τεράστια πίεση. Και τα τελευταία στοιχεία της 1ης Οκτωβρίου λέει 24% ε, ποσοστό πληρωμής αλλά οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι 350%. Οπότε, ερωτώ, αν η πίεση είναι υψηλή, οι τράπεζες θα θαθανίσουν και οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα μπορούν να σε χρηματοδοτήσουν. Τι θα προτείνετε εσείς, αύξηση των προκαταβολών ή επαναφορά μιας πρότασης που απέρισε το Συμβούλιο για δύο χρόνια να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αύξηση της χρηματοδότησης που δεν μπορούν να αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Αυτό που λέμε decommitment έχει διτή μορφή. Απ' τη μία επιβάλλει πειθαρχία, απ' την άλλη δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πλήρη κατάργηση της χρηματοδότησης, Υπάρχει δηλωμένη βούληση του Συμβουλίου, οπότε θα είναι αδύνατο κάτι τέτοιο. Αποκλείεται να επαναληφθεί αυτή η πρόταση. Καλύτερα να επικεντρωθούμε στις ε, αυξημένες προκαταβολές και άλλες προφυλάξεις που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο γύρους. Ο πρώτος γύρος έγινε το 2008 και ο δεύτερος το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των ε, κονδύλιων συνοχής. Ακριβώς για να αντιμετωπίσει την κρίση. Θα επικεντρωθούμε στο ότι είναι εφικτό και πολιτικός αποδεκτό. Σας ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, στο μέτρο που ο κοινοτικό προπολογισμό χρηματοδοτείται με τον τρόπο που, που χρηματοδοτείται, είναι σαν να, ε, να δαγκάνει ο σκύλο στην ουρά του. Γιατί τους άλλους τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούν τον κοινοτικό προπολογισμό. Το θέμα είναι πώς θα γίνει η χρηματοδότηση από τον εθνικό προϋπολογισμό ή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και αυτό είναι από πολιτική άποψη πολύ σημαντικό το θέμα. Ένα μικρό διάλειμμα τώρα με παρεμβάσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Περιφερειακής που ζήτησαν το λόγο για να θέσουν ερωτήσεις. Καλωσορίζω τον πρόεδρο Τεκάστρο που εκπροσωπεί την Επιτροπή Γεωργίας και δικαιούται πέντε λεπτά, λυπούμε μου που έχετε τόσο λίγο χρόνο για να θέσετε τις ερωτήσεις Μονόλεπτη ερώτηση του Πρόεδρου Δεκάστρο, δίλεπτη απάντηση του προτινόμενου Επιτρόπου και δυνατότητα δευτερολογίας μονόλεπτη για τον κύριο Δεκάστρο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μασούρ και σας ευχαριστώ και εκ μέρους Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Η συζήτηση για το μελλοντικό κοινοτικό προπολογισμό ε, επηρεάζει και την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Και περιλαμβάνει τη δυνατότητα σημαντικών περικοπών των πόρων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν και σε κάποια ανεπίσημα έγγραφα που μοιράστηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Η πιθανότητα βέβαια περικοπής των γεωργικών δαπανών έρχεται σε αντίφαση με την ανάγκη ε, μεγαλύτερη συνεισφορά στις γεωργίες ό,τι αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την περιβαλλοντική ασφάλεια. Από αυτή την άποψη θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η γαλακτοκομική κρίση έδειξε ότι χωρίς παρέμβαση της κοινή γεωργικής πολιτικής θα δαπανίσουμε πολύ περισσότερα. Είδαμε τις παρεμβάσεις Γαλλίας, Ισπανίας και Γερμανίας και θα δημιουργήσουμε όλο και μεγαλύτερες στρεβλώσεις στην κοινή εσωτερική αγορά. Στι Ηνωμένε Πολιτείες πέρυσι αυξήθηκαν οι γεωργικέ δαπάνες και το 2009 ξεπέρασαν τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Κυρίως ε, χάρη στην αύξηση των πόρων για τις αντισυγκυριακέ ε, πληρωμές και τα εθνικά προγράμματα επισητιστική ε, αρρωγής. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε 2 εκατομμύρια γεωργούς ε, στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 10 εκατομμύρια γεωργούς. Ποιες είναι οι απόψεις για τα μελλοντικά κονδύλια που θα πρέπει να αφιερωθούν στην κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει στη γεωργία τη λιγότερο από το 1% των συνολικών δημοσίων δαπανών τη. Πολύ λιγότερο δηλαδή από αυτά που δαπανούν οι Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν λιγότερου γεωργού. Ευχαριστώ για δύο λεπτά ο κύριο Λεβαντόφσκι. Δίκιο έχετε κύριε Πρόεδρε ότι σε αντίθεση με την ε, γνώμη του κοινού οι γεωρικές δαπάνες είναι λιγότερο από 1% του ΑΕΠ, του συνολικού ΑΕΠ. Ούτε καν μισό εκατό του ΑΕΠ. Γιατί είναι αμυγός κοινοτική αυτή η πολιτική. Και υπάρχουν βέβαια μερικές διαφορές μεταξύ των νέων κρατών μελών για τις άμεσες πληρωμές. Υπάρχει μία εξέλιξη, γιατί στη δεκαετία του 80 κατανάλωνε πάνω από το 70% του κοινοτικού προπολογισμού, ενώ στο τέλος των δικών μας δημοσιονομικών προοπτικών απορροφά το 30 με 35%. Αλλά γίνεται ένα είδος προμαγειρέματος, προτιγανίσματος της γεωρικής πολιτικής, όπως έγινε το 2002. Προγραμματίζουμε τότε τι ε, δημοσιονομικε προοπτικε προοπτικές 2007-2013, η περίφημη Συμφωνία Γερμανία για το μέλλον. Αυτό το είδο του προμαγειρέματο ε, φαίνεται ότι γίνεται και τώρα. Γιατί στην πρωτεύουσα της πατρίδας του Αλάου γίνονται κάποιες συναντήσεις ε, Υπουργών Γεωργίας και η πλειοψηφία των Υπουργών Γεωργίας έχει κοινή θέση. Φαίνεται ότι το γεωργικό λόμπι είναι πολύ καλά οργανωμένο στην Ευρώπη, σε αντίθεση πάλι με το λέγω αίσθημα και με την κοινή γνώμη. Γιατί πάνω από 20%, πάνω από 20 υπουργοί γεωργίας είναι υπέρ τη συνέχισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Υπάρχει μία σύμπνη. Άλλωστε το γεωργικό μοντέλο είναι ένα απόσπαστο τμήμα του ευρωπαϊκού μοντέλου ζωή. Γιατί να το τροποποιήσουμε. Είπαμε θα αλλάξει κάπως με την πολλαπλή συμμόρφωση για παράδειγμα, το cross compliance, προκειμένου να λάβει υπόψη ε, και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων. Το θέμα της διαφοροποίησης, του modulation, ίσως αποτελέσει τμήμα μιας μελλοντική γεωργικής συμφωνίας, αλλά μου είναι αδιανόητο να επαναθηνικοποιήσουμε ή να καταργήσουμε ολοκληρωτικά αυτό το σημαντικό τομέα των κοινοτικών μας προσπαθειών προσπαθειών που γίνονται φυσικά και από δημοσιονομική άποψη. Σας ευχαριστώ. Θέλετε και πάλι το λόγο κύριε Πρόεδρε. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για την απάντηση κύριε Επίτροπε. Και με βάση αυτά που είπατε στο τέλος σας ερωτώ. Συμφωνείτε ότι η επανεθνικοποίηση της γεωρικής πολιτικής θα επιφέρει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε, Σας ευχαριστώ, κύριε ναι, η απάντηση είναι ναι. Και αυτό ήταν από τα επιχειρήματα στην διαμάχη κατά της επανεθνικοποίησης. Είναι πολύ το θέμα της χρηματοδότησης της γεωργίας και της ε, πολιτικής συνοχής. Είναι το πολιτικό θέμα <clears throat> του ενός προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης κατά πόσο θα πρέπει να είναι θέμα γεωγραφικής συνοχής όπως ήταν πριν από τις δημοσιονομικές βλέψεις. Μέσα στα πλαίσια του δεύτερου κεφαλαίου της γεωργικής πολιτικής. Διαφοροποίηση, ναι. Εθνικοποίηση, έχω ενδιασμούς. Πρώτα σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε τον πρόεδρο Τεκάστρο για την παρουσία του και τις ερωτήσεις του. Η κυρία Χίμπνερ, το μεταξύ που είναι πρόεδρος της περιφερειακής Πολιτικής, είναι εδώ μαζί μας. Τι χαιρετίζω και όπως και ο κύριος Δεκάστρο έχει δικαίωμα. Ένα λεπτό, λυπούμε. Ένα λεπτό μόνο, κύριε πρόεδρε. Και μετά θα μπορέσετε να ξαναπάρετε το λόγο και ένα λεπτό μετά την απάντηση στην ερώτηση που δώσε ο κύριος Λεβαντόσκη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα σα υποβάλω την ερώτησή μου στα αγγλικά. Στην γραπτή σας απάντηση στο ερώτημα υπ. 4 λέτε ότι είναι απαραίτητο να εστιαστεί ο μελλοντικό προπολογισμό εκεί που υπάρχουν πραγματικές προκλήσεις, ανταγωνιστικότητα, κλιματολογικές αλλαγές και ενέργεια. Και σίγουρα ξέρετε ότι η μεταρρύθμιση της συνοχής ε, το 2006 επανεξτίασε την πολιτική αυτή ακριβώς το θέμα αυτό ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, κλιματολογικές ε, αλλαγές, ενέργεια, αποτελεσματικότητα. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν πολύ σύντομη και θα σας ήμουν ευγνώμη να μου εξηγήσετε γιατί δίνετε την εντύπωση ότι θεωρείτε ότι οι παραδοσιακές πολιτικές δεν δίνουν απαντήσεις στις μελλοντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ κ. Λεβαντόφσκι. Ναι, μιλάμε μεταξύ μας, αλλά στα αγγλικά. Καλά. Ε, δεν είναι απόλυτα σωστό. Γιατί και στην εισαγωγή μου είπα ότι δεν είναι ξεπερασμένο κάθε τι το παραδοσιακό, αλλά προσπαθούμε να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ καινοτομία και ε, της σοφίας των παλιών διακανονισμών. Και ε, ξέρουμε ότι και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φτάνει μέχρι το τοπικό επίπεδο. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που το μάθαμε στην πράξη με τις επιτροπές μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εδώ έχουμε μία μεταφορά κέντρου βάρου στην αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής ε, που θα πρέπει να είναι σύμμορφη με αυτό που σας προανέφερα. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των περιφερειών, όχι μόνο να ξεπεράσουμε κάποια όρια, αλλά να ξεπεράσουμε τις ιδέες. Αυτή η αλλαγή παραδείγματο οδηγεί στο να εξετάσει τώρα η συνοχή σαν μια δυνατότητα ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, πράσινης οικονομίας που εν μέρει έχουν συμμεληφθεί μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης λισαβονοποίηση ε, της πολιτικής συνοχής. Δεν είμαστε εδώ αντίθετοι με την έδεια της ε, περιφερειακής συνοχής όπως αναφέρεται στη συμφωνία στην, ε, της ε, Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ε, είμαι πολύ ευγνώμων προς εμάς για τις ιδέες σας που φαίνεται ότι διαφορούν με αυτό που ε, θεωρούσε Θεωρείτε ότι η πολιτική συνοχή είναι μια σύγχρονη πολιτική. Σας ε, παρακαλώ το έχετε κατά νου αυτό όταν διευκολύνετε την προσαρμογή και την προετοιμασία των νέων δημοσιονομικών προβλέψεων. Θα ήθελε κύριε μέλλον ε, επίτροπε να ξέρετε ότι οι ιδέες που θα έχουμε μέσα στα πλαίσια και των κλιματολογικών αλλαγών και της καινοτομίας απαιτούν ακριβώς στον τομέα αυτό δράση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επανερχόμαστε τώρα στα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών και θα ήθελα να δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Χωσή Μανουέλ Φερνάς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε την αλληλεγγύη της, δεν ξέχασε τους άλλους και απόδειξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς καν διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει ε, ε, εξουσίες για το θέμα αυτό, πρόβλεψε ένα ειδικό ταμείο ε, μέχρι το 2012 για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ταμείο, ε, να βοηθούμε τους άλλους, αλλά να μην ξεχνούμε και τους εαυτούς μας. Ερωτώ λοιπόν, δεν θεωρείτε ότι ήδη από τώρα σε θέματα επιστημονικής έρευνας και σε θέματα πειραματικών προγραμμάτων και πιλωτικών σχεδίων θα πρέπει η Ευρώπη, τα κράτη-μέλη της, για να μην χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να συνδυάσουν την ανταγωνιστικότητα με τη φιλοδοξία τους να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει ήδη από τώρα να επενδύσουν και να ενισχύσουν τα σχετικά προγράμματα μια και ήδη μια τέτοια επένδυση θα πρέπει να έχει αντίκτυπο και στο πολιτέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ για δύο λεπτά, κύριο Λεβαντόφσκι. Η έρευνα και οι δημόσιες δαπάνες στην έρευνα δίνουν την εντύπωση ότι εδώ έχουμε εμπορικά πρότυπα και βελτιώσεις. Όχι έναν αυτό σκοπό. Δεν είναι αυτό σκοπός ε, οι δαπάνες. Θα πρέπει κατόπιν να υπάρχει ένα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο αποτέλεσμα. Και ε, όσον αφορά τις προτάσεις των δημοσίων δαπανών για την έρευνα, δεν έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση εδώ σχετικά με άλλες χώρες. Αυτό που μας λείπει είναι ε, το στοιχείο του ιδιωτικού τομέα που ήταν σαφές ε, με την αποτυχία του Γαλιλαίου που καταρχήν θεωρήθηκε μια εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και τώρα έχουμε μόνο δαπάνες δημοσίου χρήματος Πράγμα που μας κάνει να προβληματιζόμαστε και σχετικά με μελλοντικού προπολογισμού. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της έρευνα και όχι όσον αφορά μόνο το ύψος των κονδυλίων, αλλά και με την ε, παράδοση στις επιχειρήσεις, το θέμα της κοινοτομίας στις επιχειρήσεις και όλες τις κοινωνικές επιπτώσεις που εμπλέκονται και που χρειάζονται ούτως ώστε το δημόσιο χρήμα να περάσει στην έρευνα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της κοινωτικής οικονομίας. Αλλά ξεκινήστε με το άλλο θέμα, το κατά πόσο θεωρούμε αυτούς υποχρεωμένοι προς τις φτωχότερες χώρες. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών που πρέπει να υπομισθούν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ε, για τις φτωχότερες χρόνες. Αυτό που πληρώνουμε εμείς από το κοινωνικό προπληρωισμό 105 εκατομμύρια για 2010-2012 είναι μικρό σχετικά το ποσό. Δευτερολογία, όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Φραντσέσκα Μπαλτσάνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε συχνά τον όρο ευελιξία. Είναι αναπόφευκτο βέβαια, γιατί ένας προπολογισμός είναι τόσο πιο αποτελεσματικός όσο πιο ευέλικτος είναι. Και το μέσο της ευελιξίας που προβλέπεται από την Διαθεσμική Συμφωνία είναι ένα μέσο ισχυρό που θα μπορούσαμε όμως να το ενδυναμώσουμε για να αντιμετωπίσει μια πρόκληση όπως την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Θα ήθελα να ξέρω πώς έχετε επιλέξει εσείς συγκεκριμένα τα πράγματα, πώς μπορείτε να δώσετε εδώ περισσότερη ευελιξία στο κοινωτικό προπολογισμό. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριο και για δύο λεπτά παρακαλώ. Αυτό ήταν μία από τις σημαντικότερες δηλώσεις που έκανα. Δεδομένων των περιορισμών θα πρέπει να έχουμε περισσότερη ευελιξία. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μέσω των μέσων που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ευελιξία που τη χρησιμοποίησαμε πολλές φορές σε διαπραγματεύσεις το παρελθόν. 90 εκατομμύρια νομίζω δόθηκαν πέρσι για ευελιξία μέσα στα πλαίσια του 2010. Αυτό που είναι καλό για το μέσο αυτό της ευελιξίας είναι ότι μπορεί να περάσει στα επόμενα έτη. Γι' αυτό το ύψος των κονδυλίων της ευελιξίας αυξάνεται και έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε το μέσο αυτό στους προπολογισμούς που θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά άγνωστα θέματα νέες υποχρεώσει, νέες δεσμεύσει που καμιά φορά εκπλήσουν το Κοινοβούλιο ή εκπλήττουν την Εκτελεστική Επιτροπή. Και ξαφνικά ζητάτε να δώσουμε χρήματα, να βρούμε νέα χρήματα. Την τελευταία, λοιπόν, ένα ε, περιθώριο ευελιξία 200 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και τα 500 εκατομμύρια από το Ταμείο ε, Πασκοδιώτες και ένα δις από το Ταμείο Λεγγύης. Αυτό μας δίνει κάποιες δυνατότητες ελιγμών μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης ε, του, της 2007 2007-2014 και μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται πέρα από αυτά. ευχαριστώ. Η Φραντσέσκα, ένα λεπτό. Pensa che sia prioritario intervenire. Είπατε ότι έχετε προτεραιότητα στις μέγιστες οροφέ των πιο προβληματικών τίτλων και κεφαλαίων, το 1α και το 4, Φερρυπίν. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Ο κύριο Λαβαντόφσκι. Έχω μπροστά μου τον πίνακα τι προβλήματα θα έχουμε τα επόμενα χρόνια και αν δείτε τον προπολογισμό του 2010 έχουμε μια καλή εικόνα. Το 1α περιθώριο 0, 1β περιθώριο 0, 3α 19 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 0. 4, 1 εκατομμύριο. Δεν έχουμε περιθώρια καθόλου. Και το ίδιο ισχύει και τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε πάρει, θα πρέπει να προχωρήσουμε με την ευελιξία. Άλλο τρόπο δεν έχουμε για την αναθεώρηση. Έχουμε κάνει πολλές αναθεωρήσεις του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό όμως δεν ήταν ένα καλό μήνυμα για τον ε, κεφάλαιο 2. Πρόεδρος, αυτή η σειρά 0-0-0 είναι μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Τώρα, το λόγο σε αυτόν που έσωσε την, ε, την συντακτική συνέλευση, το Βέλγιο, και πως μας σώσει και πάλι στον Ζακ Λίκ Ντεάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Στην απάντησή σας είπατε ότι η συνθήκη της Ρώμης έδινε διαφορετικό νόημα στους ίδιους πόρους από ό,τι δίνουμε σήμερα. Γιατί ήταν τελωνιακοί δασμοί οι οποίοι πηγαίνουν κατευθείαν στα ταμεία της Ένωσης. Τώρα έχουμε ιδίω πόρου που προέρχονται από του εθνικού προπολογισμού. Δεν είναι καλή λύση αυτή, από τα κράτη-μέλη έχουν δυσκολίε δημοσιονομικέ λόγω τη κρίση. Από τη μια μεριά έχουμε ερωτήματα μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας που δίνει περισσότερα δικαιώματα στην Ένωση. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, πάμε κάπως στραβά. Το θέμα λοιπόν των ιδίων πόρων σύντομα, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα αποκτήσει ιδιάζουσα σημασία. Θεωρώ ότι η Κομισιόν καλείται να παίξει ενεργό ρόλο. Σκοπεύετε να δράσετε ενεργά εξ ονόματος της Επιτροπής στο θέμα αυτό. Ο κύριος Λεβαντόφσκι να μας απαντήσει έχει δύο λεπτά. ήδη οι πόροι. Αμέσως έρχεται στο νου το όνομα Λέν Λαμασούρ, γιατί αυτός ξεκίνησε τη συζήτηση για την αναθεώρηση και το μέλλον των ιδίων πόρων με το έγγραφο εργασία του και τις συναντήσεις που είχε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σήμερα ήδη είπαμε ότι η διάγνωση είναι πάνω κάτω η ίδια. Δηλαδή, το ισχύον σύστημα και με τα πορίσματα του Συμβουλίου του 2005 είναι τόσο περιπλεγμένο, με ένα σωρό εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων, είναι τόσο μακριά από τη συνθήκη της Ρώμης, τόσο μακριά από την αρχική ιδέα των ιδίων πόρων, το 75% εξαρτάται από συμβολή των κυβερνήσεων. που συνδέεται με την νοοτροπία θέλω τα λεφτά μου πίσω. Το καθαρό υπόλοιπο, η καθαρή συνεισφορά. Όσον αφορά τη διάγνωση, είναι σαφής. Όσον αφορά τις προτάσεις, παραδείγματος χάρη η πρώτη ομάδα του Μπαρόσο υπήρξε παθητική όσον αφορά το θέμα των ιδιών πόρων μετά την εμπειρία της Επιτρόπου Στράγερ που έκανε τις προτάσεις, τις έβαλε στο τραπέζι. Υπήρξε μια φιλανδική πρόταση καθαρή συνεισφορά των κρατών μελών. Άλλες λύσεις αναφέρθηκαν επίσης σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Αλέν Λαμασούρ γιατί ήταν πολύ πιστικός και τώρα είναι δική μου ευθύνη να επανεργοποιήσω σε δύο φάσεις την πρώτη αναθεώρηση, στη δεύτερη νέα πρόταση. Φυσικά θα ρίξουμε στο τραπέζι μια νέα πρόταση για ιδίους πόρους που να είναι πολιτικά εφικτή, υλοποιήσιμη που θα ήθελα να έχω στο κέντρο του χαρτοφυλακίου μου αλλά είναι ουσιαστικά στα χέρια των κυβερνήσεων ακόμα. Και θα μπορούσα να αναφέρω και τον Πρωθυπουργό Μπράουν, ο οποίος πρόσφατα προσπάθησε μια νέα φορολόγηση Willow Lost America. Και τώρα το λόγο στον κύριο Στεφάν Λεφόλ. Καλημέρα κύριε Λεβαντόφσκι. Συνεχίζω στο ίδιο πνεύμα την ερώτησή μου. Απαντήσατε ως καλός διαχειριστής και γνώστης του προϋπολογισμού. Αλλά ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με το ύψος του κοινωτικού προϋπολογισμού. Έχουμε τους πόρους, τους ίδιους πόρους απαντήσατε. Ποια είναι η γνώμη σας. Λύνουμε οριστικά το θέμα με ένα μικρό Προπολογισμό της Ένωση είστε ένα επίτροπος που θα προωθήσετε έναν ισχυρό προπολογισμό για να δοθεί στην Ευρώπη η δυνατότητα να είναι πρωταγωνιστής σε θέματα βιώσιμη, ανάπτυξη, καινοτομίε, έρευνα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Και ένα σχόλιο για τα γεωργικά. Είπατε διαφοροποίηση, ε, συγκεκριμένη πολιτική, όχι επανεθνικοποίηση. Είστε υπέρ της επαναχρηματοδότησης των δύο πυλώνων της ΚΑΠ ή όχι. Πρόεδρος. Κύριε Ρεβαντόφσκι, έχετε δύο λεπτά. Ε, εφόσον έχω δημοσιονομικό χαρτοφυλάκιο, όσο πιο πολλά τόσο καλύτερα θα έλεγα. Πιο μεγάλο ο ρόλος μου. Αλλά θα πρέπει να λάβω υπόψη την πραγματικότητα. Ζούμε ακόμα κρίση στην Ευρώπη. Προσπαθώ να είμαι λοιπόν ρεαλιστής. Είχαμε την αρχική πρόταση της Κομισιόν του 2004 και το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων το 2006 για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013. Τα νούμερα είναι δεδομένα. είναι κάτι σαν τους αστερίσκους και τις τροπολογίες της αναγνώσης του Κοινοβουλίου. Έχουμε όμως μια νέα διαδικασία, όπως ξέρετε. Η ρεαλιστική λοιπόν υπόθεση για τον προϋπολογισμό είναι θα συνεχίσουμε με λίγους πόρους και όλο και πιο πολλές ανάγκες. Παράδοξο αυτό. Περισσότερη Ευρώπη θα πρέπει και περισσότερα χρήματα. Έχουμε την τιμαριθμοποίηση του προπολογισμού. Οι προπολογισμοί αυξάνονται. Αλλά οι δημόσιες δαπάνες, ακόμα και χωρίς την κρίση και με τα πακέτα τόνωσης, μεγαλώνουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή οι δημόσιες δαπάνες, οι κρατικοί προπολογισμοί αυξάνονται πιο γρήγορα από τον κυρωτικό προπολογισμό, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και εκεί έγινε το πρόβλημα είναι ευκολότερο να περιορίσουμε την συνεισφορά στον κοινωτικό προπολογισμό από ό,τι στον εθνικό προπολογισμό. Γιατί μετράει η δημοκρατική κοινή γνώμη σε κάθε χώρα μέλος. Γι' αυτό θέλω να είμαι ρεαλιστής. Πρόεδρος, ο κύριος Λεφόλ, δευτερολογία, ερώτηση. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε περισσότερο με τους πρωθυπουργούς για να είστε ρεαλιστής ή θέλετε να είστε φιλόδοξος τεσόμενος με το Ευρωκοινοβούλιο. Απλή η ερώτηση κύριε και απαντήσει. Αν είναι απλή δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε, θα το δούμε στην πράξη. Εγώ προσπαθώ να είμαι ένας μεσολαβητής. Θα προτιμούσα να έχω περισσότερα χρήματα, γιατί βλέπω τις προκλήσεις. Τεράστιες είναι. Πέραν του κλίματος, έχουμε τεράστιο πρόβλημα για την χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, του Γαλιλαίου και των μεγάλων προγραμμάτων που απαιτούν δις ευρώ, δις. Είναι απρακτικό τεστ όμως αυτό. Εγώ σας είπα θα είμαι ρεαλιστής. Προέρχομαι από χώρα συνοχής. Προέρχομαι από μια χώρα που είναι ο, ο πιο μεγάλος ωφελούμενος από τις, κοινωνικές, από τις κοινωτικές δαπάνες. Αλλά από εθνικοποίησα κάπως τον εαυτό μου. Πρόεδρος, άρα εμείς θα αποφασίσουμε αν όποιος δεν είναι με μας είναι εναντίον μας ή αν όποιος δεν είναι με μας είναι με μας. Που δεν είναι εναντίον μας μάλλον είναι με μας. Εμείς θα το αποφασίσουμε. Συνεχίζουμε. ήρθε καθυστερημένα λόγω κλιματολογικών συνθήκων δύο μέλη που θα πρέπει να μιλήσουν στην αρχή. Η κυρία Αντρεάσεν, εξ ονόματος της ομάδας EFD. Μία ερώτηση, ένα λεπτό. Ο κύριος Λεβαντόφσκι απαντά δύο λεπτά και αν θέλει μπορεί να δευτερολογήσει. Αντρεάσεν. Euh, euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που ήρθα καθυστερημένη. Είχα δύσκολη πρόσβαση στις Βρυξέλλες. Ερώτηση. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια ο προπολογισμό της Ένωσης δεν δαπανήθηκε 100% στο τέλος του οικονομικού έτους. 10 με 15% παραμένει χωρίς να έχει δαπανηθεί. Κατά την άποψή μου, αυτό μας δείχνει ότι δεν γίνεται σωστή ανάλυση και διαβούλευση στην προετοιμασία του. Τα αιτήματα θα πρέπει να έρχονται από τις χώρες μέλη. Το ότι οι κανονισμοί είναι περίπλοκοι δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την διαδικασία προγραμματισμού. Πρώτη ερώτησή μου λοιπόν, πώς σκοπεύετε να οργανώσετε τη σύνταξη του προπολογισμού και την προγραμματική δουλειά για τα επόμενα χρόνια. Δεύτερη ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν είχε τη δυνατότητα να αυξήσει το επίπεδο δαπανών στις διάφορες γραμμές, επ' αυτού, ποια θα ήταν η άποψή σας. Απάντηση. Ευχαριστώ. Δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Το ένα είναι οι, οι και τι δεν έχει δαπανηθεί αυτό οφείλεται στο ότι από τη μια μεριά έχουμε πληρωμέ που πάνε πέραν των δημοσιονομικών προοπτικών, από την άλλη μεριά έχουμε τι ε, υποχρεώσει. Υπάρχουν πάρα πολλέ υποχρεώσει, πάνω από 150 δι ευρώ. Και το θέμα είναι πώς συνδέονται αυτά με διαχειρίσιμο τρόπο μεταξύ των πληρωμών και των υποχρεώσεων. Πάντα θα υπάρχει αυτή η διαφορά. Το δεύτερο είναι χρήματα που δεν δαπανήθηκαν που είναι φιάσκο της πολιτικής. Δεν μιλάμε για λάθος εδώ, είναι άλλο θέμα αυτό. Χρήματα που έχουν δεσμευτεί σε μερικές περιπτώσεις ήταν ένα φιάσκο επειδή δόθηκαν τα χρήματα σε μια πολιτική αλλά δεν εκτελέστηκε η πολιτική αυτή. Οι λόγοι έχουν συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Τώρα, αν λύση θα είναι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που να διευκολύνει γνωρίζετε καλύτερα από μένα γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο πώς εξυγχρονίζεται ένας δημοσιονομικός κανονισμός έτσι ώστε να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία και να έχουμε λιγότερο ποσοστό μη δαπανηθέντων χρημάτων. Όσον αφορά δε τον προγραμματισμό, θα δούμε ποια είναι η αιτήσια ε, στρατηγική. Έχει καθυστερήσει κάπως η Επιτροπή όπως βλέπετε, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουμε ένα πρώτο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πριν από αυτόν είχαμε την αιτήσια στρατηγική. Φέτος έχουμε καθυστερήσει αρκετά, αλλά είμαστε στην αρχή ενός κύκλου. Είμαστε στην αρχή ενός κύκλου προγραμματισμού. Η κυρία Αντρεάσεν. Δευτερολογία. Σας ρώτησα ποια είναι η γνώμη σας αν θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αυξήσει ορισμένα κονδύλια. Απάντηση έχουμε συναπόφαση. Τώρα καλείται η τακτική νομοθετική διαδικασία. Δεν μπορεί μονόπλευρα να αλλάξει τον προπολογισμό. Χρειάζεται συνένωση των δύο βραχιώνων της δημοσιονομικής αρχής. Και είναι εύκολο να βρεθεί ε, να υπάρξει μια πρόταση αύξησης εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου, πιο εύκολο να γίνει αυτό παρά να το δεχτεί το Συμβούλιο. Πολλέ φορέ το Συμβούλιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών με του δικού του υπολογισμού, γιατί αυτή είναι υπεύθυνη για τι εθνικέ εισφορέ, τα χρήματα που θα πάνε στι περιφέρειε. Άλλου υπολογισμού κάνουν λοιπόν οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτό είναι πέραν των εξουσιών του Κοινοβουλίου, ακόμα και με τη νέα συνθήκη δεν μπορεί μονόπλευρα να επιφέρει αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βέρτμαν, εκ μέρου των μη εγγεγραμμένων, για ένα λεπτό. Äh, Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήρθα καθυστερημένα. Δυστυχώ αυτό λόγω των καιρικών συνθητών. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία αφορά το Ταμείο Παγκόσμιου Πίση. Πώ θα εξασφαλίσετε ότι τα χρήματα φτάνουν πραγματικά στου ενδιαφερόμενου. Δηλαδή δεν θα πρέπει να το δώσουμε στα κράτη, αλλά εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ θα ελέγξουμε ότι φτάνουν στου δικαιούχου. Και το δεύτερο ερώτηση αναφέρεται στην πολιτική κτηρίων. Ήδη θίγει το θέμα, αλλά θα ήθελα να ξέρω η συνοχή της πολιτικής αυτής κτηρίων πώς θα συγκεκριμενοποιηθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεβαντόφσκι. το θέμα της παγκοσμιοποίησης και της κτηριακής πολιτικής κάπως το αναφέραμε και προηγουμένως. Για την παγκοσμιοποίηση έχουμε έναν μηχανισμό δεν μπορούμε να τον αφισβητήσουμε ούτε αυτόν ούτε τους κανόνες του παιχνιδιού. Απλώς μπορούμε να εξακριβώσουμε αν εφαρμόζονται και να τους τροποποιήσουμε αυτούς τους κανόνες. Αυτό δεν είναι το θέμα όμως της ε, διοργανικής συμφωνίας ή της προηγούμενης. Χρειαζόμαστε πιο διεξοδικές και εμβριθείς συζητήσει. Δεν θα υπερτιμούσε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Εκτιμώ όλες τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του κατοφλίου και την αύξηση της διαθεσιμότητας των κονδυλίων παγκοσμιοποίησης ε, του 2009, ώστε να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση. Γιατί τώρα έχουμε το κατόφλι στα 500 και όχι στα 1000 όπως αρχικά. Είναι ένας χρήσιμος μηχανισμός για να γίνει πιο ελαστική χρήση των πενιχρών πόρων που έχουμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολλές ανάγκες, ιδιαίτερα και από τη μετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων. Εκτός από το Βατικανό, νομίζω ότι είμαστε η μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο ε, μεγαλύτερη χώρα ή μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος οργανισμός που κατέχει ακίνητα. Έχουμε τόσους οργανισμούς, τόσα γραφεία και πολλαπλή εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλά αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά όλα αυτά δεν αρκούν. Και απάντησα έτσι και στην ε, κυρία Χολμάιστερ. Έχουμε μια πολύ ε, φιλόδοξη και διορατική πολιτική για την πολιτική ακινήτων. Δευτερολόγια δεν υπάρχει, οπότε δίνω το λόγο στην Ingeborg Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ, σαν συνήθεια, για τον ε, προπολογισμό. Μου κάνει εντύπωση ο μεγάλος αριθμός των διατάξεων που πρέπει να τηρηθούν στο Ευρωπαϊκό ε, Ελεκτικό Συνέδριο υπάρχει ένα κείμενο με μια μισή σελίδα μόνο των διατάξεων. Εσείς προτίθεστε να ζητήσετε να γίνει μια ένωση των, ε, των ε, εγγράφων αυτών. Τώρα λέτε ότι θα είσαστε ένα honest broker, ένας τίμιος διαμεσολαβητής. Πόσο τίμιος είναι ο μεσολαβητής αυτός τι θα γίνει με την εξωτερική υπηρεσία που δεν έχουμε ακόμα καμία ιδέα για το πώς θα διαβεβαιωθεί. Γιατί η Κομισιόν δεν προσπαθεί να έχει σύμμαχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, να επιμείνει σε κοινά σημεία και γιατί η Κομισιόν δεν ρωτάει τους δικούς τους εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό που μέχρι στιγμής έχουν μείνει εκτός νυμφώνος όσον αφορά την προετοιμασία της υπηρεσίας. Ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι. Γκρέσλε είναι, έχει αναφυσβήτητο κύρος και αυθεντία για τα θέματα αυτά και είναι σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε συζήτηση αναθεώρησης ή ιστορίας του δημοσιονομικού κανονισμού. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε πολύ περισσότερο στις αναθεωρήσεις του 2006 ενώ τώρα έχουμε συναπόφαση και στο μέλλον ο δημοσιονομικός κανονισμός εμπίπτει στη διαδικασία της συναπόφασης. Δεν είμαι ακόμη έτοιμο να απαντήσω στην πρώτη σα ερώτηση. Και μάλιστα και πριν την ακρόαση, με συμβούλευσε να πω τουλάχιστον μια φορά ότι δεν είμαι έτοιμο να απαντήσω. Ε, δράτω με τι ευκαιρίε να χρησιμοποιήσω τώρα ε, αυτό το χαρτί του ότι δεν είμαι έτοιμο. Σε ό,τι αφορά τον αμερόληπτο διαμεσολαβητή, τον έντιμο διαμεσολαβητή και την εντιμότητά του, ε, δώστε μου μια ευκαιρία. Δώστε μου μια ευκαιρία να το αποδείξω μην δοκιμάζετε την καλή μου θέληση σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που δεν καλύπτει όμως όλη την ιστορία των δημοσιονομικών θεμάτων για το κατά πόσο θα εφαρμοστεί το στοιχείο του fast track της ε, α, γρήγορης ε, ταχείας διαδικασίας ή όχι. Όταν ε, ετοίμαζα την ακρόαση, μας προειδοποίησαν με την κυρία Άστον ότι από την πρώτη ώρα την πρώτη ακρό... της πρώτης ίσως ε, εμπλακούμε σε διαξυφισμούς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμα γιατί αν χρειαστούμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης στα τέλη Απριλίου θα είναι fast track διαδικασία. Ταχεία. Τώρα, αν δούμε τη διατύπωση του σημείου 17 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βλέπετε ότι είναι αρκετά ελαστική. Δεν λέει «σώνει και καλά να γίνουν όλα στα πλαίσια της τριετούς αναθεώρησης. Αλλά σίγουρα εσείς είστε ο κεντρικός, ο βασικός παίκτη. Και σίγουρα όταν εξετάσουμε τέτοια θέματα, το δικό σας όνομα, κυρία Γκρέσλε, αναφέρεται περισσότερο. Νομίζω ότι είναι πλήρως ικανοποιημένη από την απάντησή σας η Ίγκεμπορκ. Ο Λάζλο Σούριαν. úrnak például hogy rögtön a nyelvi sok... Κύριε Επιτροπέ, δεδομένου ότι έχετε πάρει θέση υπέρ της ε, χρήσης της μητρικής γλώσσας όπως κάνετε στην εισαγωγή σας, στην αρχή. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι το ένα σκέλος της αρχής του προπολογισμού και θα να ασκεί σωστά αυτή την εξουσία που έχει. Και έχουμε και μεγάλες προκλήσεις όπως πολιτική για το κλίμα, τα κοινωνικά θέματα, η οικονομική κρίση. Για πολλά από αυτά όμως την κύρια ευθύνη την έχουν τα κράτη-μέλη. Εμείς λέμε στην κοινοβουλευτική μας δραστηριότητα πολλά κεφάλαια υποχρηματοδοτούνται. Όπως οι δαπάνες για τη γεωργική πολιτική, για τη συνοχή, με μείωση των δαπανών για τη συνοχή θα βρεθούμε σε καταστάσεις όπου θα έχουμε τεράστιες διαφορές από μία περιοχή, σχέση, μία περιοχή με μία άλλη. Σχόλιο. Ναι. Ήταν πρόσφατη εμπειρία που είχαμε με την διαπραγμάτευση του προϋπολογισμού του 2010 για τα περιθώρια και τις δυνατότητες. Και εσείς ε, ξέρετε ότι προσπάθησα και εγώ ως υπέρμαχος πολυγλωσσίας ε, να δώσω μια ευκαιρία και στα πολωνικά. Δεν διήρκησε παραπάνω από ένα λεπτό όμως, γιατί όπως είπαμε και ρεαλιστή και θέλω να διευκολύνω την επικοινωνία μεταξύ μας ε, την πιο άμεση. Και αν δεν κάνω λάθος, μου θέσετε μια ερώτηση που αφορούσε το σημείο 15-16 την ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους για τη χρήση μιας γλώσσας. Παρόλο που θέλετε να αντιμετωπίσετε όλες τις γλώσσες ισότιμα. Είστε εισηγητής του θέματος αυτού και γνωρίζετε ε, ότι εκτός από το κεφάλαιο 5, βασική ζώνη ασφαλείας ήταν η γεωρική πολιτική. Αλλά το θέμα είναι να χρηματοδοτήσουμε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης. Αυτό ήταν η κύρια προτεραιότητα του προπολογισμού του 2010. Αυτό σε μεγάλο βαθμό, πέραν των άμεσων πληρωμών, δεν είναι τόσο προβλέψιμο. Δεν είναι τόσο προβλέψιμος τρόπος δρομολόγηση κονδυλίων σε ό,τι αφορά την παρέμβαση τη αγορά. Και είχαμε μερικά θετικά παραδείγματα Βέβαια τώρα η κρίση προχωρεί, αλλά όταν διαπραγματευόμαστε το προεπλογισμό το 2010 η κατάσταση πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Προσοχή λοιπόν όταν μιλούμε για περικοπές στις γερικές δαπάνες. Γιατί η γεωργική πολιτική στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό και σε παρέμβαση στην αγορά και η, η γεωργική αγορά για μένα είναι αρκετά δυσνόητη. Απέχει πόρο από το νεοκλασικό μοντέλο της οικονομικής θεωρίας. Γι' αυτό και δεν είναι και τόσο προβλέψιμη η εξέλιξη στη γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Γεντζογεύσκα. Η ερώτηση μου αφορά το κοινοτικό προϋπολογισμό του 2011. μιλήσατε για τις μελλοντικέ προκλήσεις. Εγώ βλέπω κάποιες ε, διαδικαστικές προκλήσεις, γιατί ο προϋπολογισμός του 2011 θα είναι ο πρώτος κοινοτικός προϋπολογισμός που θα εγκριθεί με βάση τις ε, διατάξεις της Συνθήκης Λισαβόνας. Κατά τη γνώμη μου σημαντικό θα είναι το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταπεξέλθει στι προσδοκίε τη χρηματοδότηση τη εξωτερική πολιτική, τη πολιτική ενεργειακή ασφάλεια με διασταλτική έννοια, πώς θα καταφέρει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα μέσα της για να χρηματοδοτήσει την ε, πολιτική συνοχής και τέλος πώς ο προϋπολογισμός του 2011 θα χρηματοδοτήσει τις δεσμεύσεις των κοινοτικών ε, οργάνων απέναντι στους υπαλλήλους και τους εργαζομένους. Επίσης, ε, το, το προσχέδιο προϋπολογισμού, πώς το αντιλαμβάνεστε. Γιατί αυτό το προσχέδιο προπολογισμού θα δημοσιευθεί εντός λίγο Και ευελπιστώ ότι θα δημοσιευθεί επί της δικής σας θητείας. Ευχαριστώ κύριο Λεβαντόφσκι. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια διαδικασία και φυσικά δεν έχουμε περάσει ακόμη στη δεύτερη φάση της διαδικασίας για το προσχέδιο. Πρώτα θα πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, θα προσπαθήσουμε να το σεβαστούμε, αλλά χρειαζόμαστε συμφωνία τον Απρίλιο στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή και για τα άλλα θέματα που είναι συναφή με τη Λισαβόνα, προκειμένου να εφαρμόσουμε εύρυθμα και απρόσκοπτα τη δημοσιονομική διαδικασία. Το δεύτερο θέμα είναι το περιεχόμενο, η ουσία του προπολογισμού. Ίσως υπάρξουν κάποιες απρόβλεπτες παρεμβάσεις στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής, αλλά πέραν αυτών έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα 75 εκατομμύρια για το κοσυφοπαίδιο, στο decommissioning. Ήταν αρκετά διεισδυτικό θέμα για το 2010 και άλλα 75 απαιτούνται για το 2011. Θα πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για το περιβάλλον. Έχουμε τον Κοπέρνικο και υπάρχουν και κάποια στάθμιτη παράγοντες, μάλλον άγνωστοι παράγοντες για άλλα προγράμματα. Οπότε αυτό θα είναι το περιεχόμενο ενός προσχεδίου προϋπολογισμού που ήδη άρχισε και καταρτίζεται αλλά με βάση κάποιες ε, προσωρινές διαδικαστικές αποφάσεις. Και μετά θα έχουμε τον κανονισμό ή μάλλον τη συμφωνία που θα μετατραπεί από το soft law των διακηρύξεων στο ουσιαστικό δίκαιο, το δευτερογενές δίκαιο για τα θεσμικά όργανα. Και σας ανέφερα λίγες μόνο από τις πολυάριθμες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2011. Τώρα για την ε, ΚΕΠΑ, ξέρετε πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα, για τα αποθεματικά, ε, εντάξει, το τέλος πλησιάζω, αυτό είναι το τελευταίο που θα πω. Τώρα υπάρχει συναπόφαση και για τα αποθεματικά και αυτή είναι σημαντική η καινοτομία. Συναπόφαση για τα αποθεματικά. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος του καταλόγου των εγγεγραμμένων ομιλητών. Καταπληκτικά τηρήσαμε τις προθεσμίες μας και το χρόνο συζήτησης. Ευχαριστώ στους αδελφούς του ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές έχουν δικαίωμα για ένα λεπτό ο καθένας. Μια συμπληρωματική ερώτηση στην οποία θα απαντήσει ο κύριος Λεβοντός με ένα λεπτό θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Βάγκα. Ένα λεπτό. Και ο κύριος Λεβοντός ένα λεπτό για την απάντηση μετά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Χούβερ αναφέρθηκε στις ανησυχίες για τις πρόσφατες προτάσεις για την πολιτική της Κομισιόν για το 2013. Θα μας πείτε πώς θα πείσετε τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση Προεπολογισμού και τους συναδέλφους στο Συμβούλιο ότι δεν θα πρέπει να ξαναεπανεθνικοποιήσουν την πολιτική αυτή του 2013. Θα υπάρχουν βέβαια και άλλα έκρεμα θέματα, αλλά είχαμε δεχθεί προηγουμένως όπως είπατε, ότι χρειαστεί κάποια αναθεώρηση των δημοσιονομικών προβλέψεων. Συμφωνείτε ότι η αναθεώρηση αυτή, αν λάβει χώρα, θα πρέπει όχι να συμπληρώνει μόνο τα όρια κάθε κεφαλαίου, αλλά να αναφερθεί και σε κάποιες αλλαγές προτεραιοτήτων και να υπάρχουν κάποιες κινήσεις μεταξύ των διαφόρων κεφαλαίων. Ευχαριστώ κύριε Λεβαντάφσκι. Ε, θα πρέπει να φτάσουμε αυτά τα μη έγγραφα τώρα. Έχουμε μία συνέχεια, έχουμε μία ανταλλαγή απόψε μεταξύ της κυρίας Σιούμπνερ και του Προέδρου Μπαρόσο. Κάποια ανταλλαγή επιστολών. Έχουμε την έγγραφα σημασία για την συνοχή. Μια πρόταση του παλαιού Επιτρόπου. Υπάρχει το θέμα αυτό της επενεθνικοποίησης. Το μόνο δε επιχείρημα που μπορώ να κατανοήσω είναι ότι αν θέλουμε να συγκεντρωθούμε στις, ε, στο να δοθεί προτεραιότητα στην πολιτική συνοχή θα μπορεί να γίνει από τον άλλο προς τα κάτω. Όχι από, το, από κάτω προς τα άνω, αλλά αυτή δεν είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι αυτό το επιχείρημα που εγώ θα χρησιμοποιήσω. Εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Αυτή τη στιγμή κανένας δεν ε, ε, εγκρίνει αυτό το μία εγγραφό, δεν θεωρεί ότι το έχει γράψει. Ευχαριστώ κύριε Λαβία. Ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Ο Επίτροπος θα αναποσίσει φαινοπέ και ο κύριος Αγγλούν επίσης ένα λεπτό. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπη, ακούσαμε να λέτε ότι δεν γνωρίζετε το περιεχόμενο του λεγόμενου non-paper, δηλαδή του εγγράφου που τυπώθηκε μεν με επικεφαλίδα της Κομισιόν αλλά δεν του αναγνωρίστηκε πατρότητα και το περιεχόμενό του δεν σας βρίσκουν σύμφωνο. Αλλά στην ακρόαση ακούσαμε επίσης να μας λέτε ότι δεν συμφωνείτε με την επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής. Συμπεραίνω λοιπόν ότι η πολιτική αυτή θα εξακολουθεί να βαρύνει και να έχει προτεραιότητα στη δράση της Ένωσης όσον αφορά τον προπολογισμό. Και σας ερωτώ, αν κατάλαβα καλά από την προηγούμενη απάντησή σας, το επίπεδο χρηματοδότησης θα πρέπει να παραμείνει εκεί που είναι. Ο κύριος Λεβαντόφσκι. Πολύ γρήγορα, Δύο λόγια για ναι, για μένα αυτό είναι ένα μη έγγραφο. Τι να σας πω, δεν υπάρχει. Για να μην υπάρχουν έγγραφο. Όσο για τη γεωργία, έχω να πω ότι αυτό έχει γίνει. Γιατί αυτή ήταν μια συμφωνία σύραξου έντερα το 2002, ότι οι προτάσεις δηλαδή της γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να κατεβεί στο 33% μέχρι το 2013. Και είχα <coughs> πει επίσης ότι κυρί, κυρίως το μης ε, του προβλησμού, το έχουμε 100% συνοχή και η Γεωργία θα πρέπει να έχουμε υπόψη στις πραγματικές εξελίξεις στον πραγματικό πολιτικό κόσμο. Και εδώ έχουμε βέβαια τις, ε, στους υπουργούς ε, συνοχής και συναντήσεις για τη συνοχή στο επίπεδο και υπουργών και στο επίπεδο παραγωγών. Λοιπόν, κάτι προμαγειρεύεται εδώ το σημαντικό αυτό του μήμα των δαπανών του προπολογισμού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριο Άκλοντ. Ένα λεπτό, <coughs> τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την ευελιξία σα για τι ερωτήσει. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο πρόγραμμα πλαίσιο για την ελληνική ανάπτυξη και μια ερώτηση που βρήθηκε προηγουμένω όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και την αξιολόγησή του που προβλέπεται μέσα στη αυτές και ε, Ε, κατά τη γνώμη σας, ποιο θα ήταν το ιδανικό χρονικό πλαίσιο για την εξέταση αυτή του προγράμματος πλαισίου υπαριθμών 7. Πότε θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η προσωρινή εξέταση και μέχρι πότε. Οπωσδήποτε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, γιατί πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική δαπάνη. από 80 εκατομμύρια συνολικά, τα 60 για το πλαίσιο έρευνας. Και εδώ πραγματικά έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί εδώ έχουμε πολλή γραφειοκρατία. Και βλέπουμε πολλά χρήματα να επιστρέφονται στις χώρες. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι να διατεθούν τα κονδύλια την έρευνα στους δικαιούχους. Αυτό είναι για μένα το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει μειωθεί. Ε, ναι. Έχει μειωθεί σε σχέση με την πρόταση Κομισιόν στο 1α κατά 20% μέσα στα πλαίσια των πραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Αλλά κατά με η έρευνα έχει σημασία για τα αποτέλεσματα, όχι για το ύψος των κονδυλίων. Και στο διευθυντικό προβλησμό για το 10 έχουμε ακριβώς μειώσω το με αυτό γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα χρήματα που διατίθενται. Αυτή είναι η απάντησή μου. Πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας παίρνουν τρία λεπτά μόνο που έχουμε στη διάθεσή μας την αίθουσα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον υποψήφιο επίτροπο που ήταν εδώ διαθέσιμο σε εμά με μεγάλη σοβαρότητα, πολλές ικανότητες και προσπάθησε πραγματικά να απαντήσει με ακρίβεια σε όλες τις ερωτήσεις και με υπομονή. Και αυτό νομίζω ότι το εκτιμήσανε όλοι οι βουλευτέ. Και θα ήθελα επίση να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω συγγνώμη, όλους τους βουλευτές της Επιτροπής Προεπολογισμών και των άλλων επιτροπών που σεβάστηκαν αυστηρά τους κανόνες και ιδίως τον χρόνο αγόρευσης. Κύριε Ρεβεντόφσκη, σας ε, υποδεχθήκαμε εδώ με ανάμεικτα συναισθήματα. Οι μεν σας ζήλευαν, προτιμούσαν ε, ίσως να είναι στη θέση σας, οι άλλοι, ιδίω οι πιο νέοι, ε, ευχόμενοι κάποια στιγμή να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Αυτό που με εντυπωσίασε στις πλούσιες αναλλαγές απόψεων που είχαμε σήμερα το απόγευμα είναι ότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουμε σύστημα. Και οι ερωτήσεις που σας υπευλήθησαν υπευλήθησαν προς ένα άτομο που θα μπορούσε να είναι επίσης υποψήφιος και για την Επίτροπος για Επιτροπή για, την, ε, για το θέμα της Γεωργίας, εξωτερικής πολιτικής, μεταφορών, ανάπτυξης, οτιδήποτε. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι στη συνθήκη της Αβώνας ο Επίτροπος για τους Προπολογισμούς θα πρέπει με στα πλαίσια του συλλογικού οργάνου της Επιτροπής, προφανώς είναι συλλογική η απόφαση πάντα, μέσα στο συλλογικό αυτό όργανο θα πρέπει να παίξει τον ρόλο του Υπουργού Οικονομικού και Οικονομίας που παίζει ένας υπουργό σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο Κράτους. Μέχρι στιγμής δεν συνέβαινε αυτό, θα είναι όμως το μέλλον. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολιτική κατάσταση και να είμαστε ρεαλιστές. Σύμφωνοι. Ταυτόχρονα όμω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κανένα μόνο ρεαλιστή, ρεαλιστής, δεν γίνεται τίποτα. Ο Ζω είχε πει τότε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα, αλλά όχι την μοιραιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα το μοιραίο στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι οι ανταλλαγέ απόψε που είχαμε σήμερα το απόγευμα καταδεικνύουν ότι υπάρχει έντονη σύγκληση πνευμάτων και ότι θέλουμε πλήρως να εκμεταλλευτούμε τις νέες αρμοδιότητες, το νέο θεσμικό πλαίσιο της συνθήκης της Αβώνα, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική κατάσταση και την οικονομική κατάσταση, χωρίς να δεχθούμε μοιριότητες και ε, να δειχθούμε ε, καινοτόμοι. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Λεβαντόφσκι.